Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καλώς ορίσατε και ελπίζω μέσα σε αυτό το χειμώνα της Σιβηρίας να βρήκατε το δρόμο σας. Εγκρίνεται η μερίσια δάταξη που έχετε μπροστά σας. Πολύ καλά σας ευχαριστώ. Έχουμε και τα πρακτικά της 26ης και της 27ης Οκτωβρίου και της 8ης Νοεμβρίου που πρέπει να εγκρίνουμε. Μπορείτε να εγκρίνετε τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο τουρισμός τώρα στην Ευρώπη. Κύριος Φιντάνζο, παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Φιντάνζο. Grazie, grazie Presidente. Iniziamo oggi questa discussione su questo importante dossier. Come tutti sappiamo il turismo è una delle Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το πολύ... σημαντικό θέμα που είναι τον, ο τουρισμός στην Ευρώπη έτσι όπως προβλέπεται, στο νέο πλαίσιο έτσι όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνης και οι ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να παρέμβουν για να μπορέσουν να επηρεάσουν τα πράγματα και να συντονίσουν δράσεις που θα έχουν ε, επιπτώσεις άμεσα στον τουρισμό. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, Επίτροπος ε, Ταγιάννη, μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της ε, ε, Λισαβόνας προέβλεψε διάφορες δράσεις. Αρχές του έτους έγινε η πρώτη συνάντηση των Υπουργών Τουρισμού που συναντήθηκαν την Μαδρίτη και ενέκριναν τη διακήρυξη της Μαδρίτης που περιλαμβάνει μία σειρά κοινών δεσμεύσεων. Στη συνέχεια έχουμε τον Ιούνιο ανακοίνωση της Επιτροπής, στην οποία παρουσιάζονται 21 δράσεις ανάπτυξης του τουρισμού στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία ανακοίνωση γενικού περιεχομένου και στην συνέχεια θα αναφέρω δύο πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Τον Οκτώβριο έγινε η σύγκληση Υπουργών Ανταγωνισμού με παρουσία των Υπουργών Τουρισμού και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις γιατί για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την επιθυμία να κάνουν επενδύσεις στον τομέα τουρισμού που είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας και θα βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση. Και οργανώθηκε εκ των υστέρων το φόρουμ στη Μάλτα όπου ο Επίτροπος Ταγιάννη παρουσίασε ένα σχέδιο με στόχο την ε, ανάπτυξη συγκεκριμένα και των 29 δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας είμαι εισηγητής επί της ουσίας, αναφέρεται σε αυτό το νέο πλαίσιο πολιτικής και στις δράσεις που προβλέπονται. Πριν να εγκριθεί η έκθεση αυτή, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε το νέο νομοθετικό πλαίσιο και ήρθα αυτή την εβδομάδα σε επαφή με τους σκιώδεις εισηγητές και τους ε, εισηγητές ε, γνωμοδοτήσεων των άλλων επιτροπών. Πρόκειται για πέντε γνωμοδοτήσεις που θα υπάρχουν για το θέμα αυτό για να μπορέσω να κάνω μία δουλειά που να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις όλων. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να έχουμε ορισμό των πολιτικών που θεωρεί το Κοινοβούλιο ότι είναι σημαντικές στα πλαίσια αυτών των 21 δράσεων και των μέσεων που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διευκρίνησης αυτών των δράσεων, έτσι όπως έκανε την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, διότι ως βιομηχανία ο τουρισμός στην Ευρώπη βοηθά την Ευρώπη να είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Θα πρέπει όμως να είμαστε ανταγωνιστικοί διότι υπάρχουν πλέον και νέες επιλογές για ε, τουριστικούς ε, προορισμούς ελκυστικούς. Θα πρέπει λοιπόν για να είμαστε ανταγωνιστικοί να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στις άλλες αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες χώρες, κυρίως τις χώρες BRIC όπως τις ονομάζουμε. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 πώς θα έχουμε επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, πώς θα έχουμε ποιοτικό τουρισμό, πώς θα έχουμε ε, ποιότητα και ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι η βάση του τουρισμού είναι πάρα πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τις οποίες θα πρέπει να βοηθήσουμε να είναι ανταγωνιστικές. Εγώ συμμερίζομαι την άποψη που εξέφρασε στην ανακοίνωσή της η ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ορίσουμε την έννοια της ε, εποχικότητας, εποχικής εργασίας και στα πλαίσια του προγράμματος Καλυψό, όπως λέγεται, να είμαστε σε θέση να δεχόμεθα και τουρίστες εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τον τουρισμό και θα επιτρέψουμε και στους πολίτες μας επιτρέψουμε στους πολίτες να ταξιδεύουν όλο το χρόνο με λογικές τιμές. Επίσης, το θέμα της αξιολόγησης των, ε, ε, του, πολιτιστικού τουρισμού και των διαφόρων ε, διαδρομών τουριστικών και προορισμών τουριστικών που έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να τονίσουμε βεβαίως και τον αηφόρο τουρισμό, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα δύο δίκτυα Eden και Ρουστούρ, τα οποία έχουμε ε, κάνει και αναπτύξει συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αηφόρο τουρισμό. Όπως ξέρετε όλα αυτά τα θέματα συζητώνται αυτή τη στιγμή και η Κομισιό θέλει να έχουμε τουρισμό ποιότητος, να έχουμε παροχή ποιοτικών ε, υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν μπορεί να ενοποιηθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά γενικότερα να προωθούμε ευρωπαϊκά πακέτα τουριστικά ποιότητας. Ένα άλλο θέμα αφορά την αηφορία και την βιωσιμότητα. Υπάρχουν πολλές ιδέες σε σχέση με το θέμα αυτό. ώστε να αναπτυχθεί ο τουρισμός βάσει αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ετικέτα ποιότητας. Αλλά βεβαίως δεν θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτού του τύπου οι ετικέτες αναγνώρισης ποιότητας. για να μην αποβούν αρνητικές αντί να είναι θετικές. Τελευταία παρατήρηση, η χρηματοδότηση. Εάν ε, είδατε τον προπολογισμό για το 2011, θα είδατε ότι τα κονδύλια που προβλέπονται για τον τουρισμό έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να οργανωθούν καλύτερα οι υπάρχοντες πόροι που υπάρχουν αλλά είναι κατακαιρματισμένοι σε διάφορες δράσεις. Επίσης, στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών 2014, 2020 θα πρέπει να δούμε το θέμα των κονδυλίων. Πρόκειται για ιδέες τις οποίες θα αναπτύξω στην έκθεσή μου και ε, θα συμπεριλάβω και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι στα πλαίσια των προτάσεων που υπέβαλε ο Επίτροπο Ταγιάννη, αλλά στα πλαίσια γενικότερα δράσεων που είναι απαραίτητε για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ε, και αναφέρομαι στην οδηγία για τα ταξίδια τα οργανωμένα για τα οποία πληρώνεται μία καταποκοπή τιμή το θέμα της χορήγησης θεώρησης επίσης και οι δυσκολίες που υπάρχουν ώρες, ώρες για κάποιες χώρες για την Κίνα, Φερρυπίνη, για άλλες χώρες. Βεβαίως, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη να μπορεί να ελέγχει τα άτομα τα οποία εισέρχονται στην επικράτειά της, αλλά θα πρέπει να δούμε μήπως βλάπτουμε με υπερβολική γραφειοκρατία πολλές φορές και τον τουρισμό που θέλουμε να βοηθήσουμε. Και βεβαίως θα αναφέρω και την πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται σε επίπεδο στατιστικών. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό για τον τουρισμό. Το περιμένει όλη η τουριστική βιομηχανία. Περιμένει όλη η τουριστική βιομηχανία τα αποτελέσματα των στατιστικών που την αφορούν. Βεβαίω σήμερα γίνεται μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, αλλά είμαι στην διάθεσή σα και στη διάθεση όλων των σχεδόν ε, συντακτών γνωμοδότηση και οποιασδήποτε επικοδομητική παρατήρηση εκ μέρου, σα Ευχαριστώ. Ε, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομικές δραστηριότητες και εν μέσω της ε, κρίσης και της ύφεση ε, και θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερο ρόλο στην ανάκαμψη και της ευρωπαϊκής οικονομίας και των εθνικών οικονομιών. Έτσι, εξαιτίας ακριβώς και της οικονομικής κρίσης, ε, αλλά και άλλων φαινομένων ανώτερης βίας που βλέπουμε ότι επενεργούν αρνητικά ε, με σαφή αντίκτυπο στον τουρισμό, ε, θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια ενιαία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, τίνοντάς τον να γίνει πιο βιώσιμος, πιο ανταγωνιστικός, ανθεκτικός και σύγχρονος. Ε, σε αυτή την προοπτική βεβαίως ο συντονισμός όλων όσων συνεμπλέκονται στην δημιουργία ε, του τουριστικού προϊόντος είναι αναγκαίος και έχει ουσιαστική σημασία η συζήτηση αυτής της έκθεσης ε, με όλα αυτά που ισχύουν μιας και ε, στην εποχή Λισαβόνας ο τουρισμός αποκτά μια άλλη διάσταση για το κοινοβούλιο μας. Όσοι ασχολούμαστε με τον τουρισμό δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε σε σημαντικά ζητήματα. Έτσι δεν θα αναφερθώ σε αυτά που ο συνάδελφος Φιντάντσα αναφέρθηκε, ε, αποσπασματικά και τηλεγραφικά ε, να αναφέρω ότι ε, ένα από τα ζητούμενά μας δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας που να εστιάζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας και που θα δώσει και τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν όλη τη βεντάλια των προϊόντων του θεματικού τουρισμού. Εδώ είμαστε εξαιρετικά συγκριτικά θετικότερη των τρίτων χωρών και θα είναι και ένα κλειδί για να ανοίξουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου που είναι κάτι που απασχολεί σχεδόν το σύνολο των τουριστικών περιοχών της Ένωσης. Νομίζω ότι η θέσπιση ενός ενιαίου προτύπου κατηγοριοποίηση των καταλημάτων θα ήταν σημαντική και θα συνέβαλε και στην προστασία του καταναλωτή αλλά και στην ποιοτική αναβάθμιση των καταλημάτων καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτές. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει την αντιμετώπιση δηλαδή μια σύγχρονη τάση δημιουργίας μονοπωλίων και ολιγοπωλίων που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά ε, και που ε, τη συναντάμε τον τελευταίο καιρό και είναι επόμενο ε, μετά την κρίση και την ύφεση να αυξάνεται είτε όσον αφορά τις εταιρείες, ε, των, τις αεροπορικές εταιρείες που βλέπουν μια τάση συγχωνεύσεων και δημιουργίας ολιγοπολίων ή την υπερσυγκέντρωση στα, στους μεγάλους tour operators ε, ιδιαίτερης ισχύω, πράγμα που δημιουργεί και προβλήματα πέραν των στρεβλώσεων της οικονομίας ε, και με τις μικρές κοινωνίες συνήθως, μιας που και η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από αυτούς τους ε, μεγάλους οργανισμούς πια, αλλά και η κατεύθυνση σημαντικού αριθμού τουριστών. Ε, νομίζω ότι μια υποκατηγορία αυτού του προβλήματος που είναι η μεθοδολογία του all-inclusive πρέπει να αντιμετωπιστεί με την έννοια της αναγκαιότητας πια θέσπισης συγκεκριμένου πλαισίου κανόνων. Να αναφέρω ε, για την αναγκαιότητα και τη διευκόλυνση που πρέπει να έχει η δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων, clusters, ε, και όσον αφορά τις ε, μικρές και μεσαίες ε, επιχειρήσεις αλλά και όσον αφορά οργανισμούς και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός πελατοκεντρικού συστήματος για την ποιοτική παρακολούθηση του ευρωπαϊκού τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος θα μπορούσε το σύστημα αυτό να βασιστεί στην ύπαρξη ενός περιφερειακού σταθμού ενός παρατηρητήριου ε, ποιότητας που θα μπορούσε να λειτουργήσει σε κάθε περιφέρεια της Ένωσης ε, με ένα κοινό λογισμικό και πληροφοριακό σύστημα για να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης των περιφερειακών τουριστικών προορισμών με βάση την άποψη και την εμπειρία του πελάτη. Θα ήταν χρήσιμο και για τον καταναλωτή αλλά και για τη λειτουργία του τουριστικού προϊόντος. Τέλος, και το μόνο που θα επαναλάβω γιατί θεωρώ ότι είναι ένα μείζον ζήτημα ε, από αυτά που είπε ο συνάδελφος Φιντάντσα είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να διευκολυνθεί η παροχή βίζας ε, σε ε, δυνητικούς επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πολύ μεγάλες καινούργιε αγορές όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία ή δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες και ίσως θα ήταν χρήσιμο να ανοιχνεύαμε τη δημιουργία κοινών προξενικών γραφείων σε τρίτες χώρες ε, που θα μπορούσε να ε, ξεπεράσει το σημαντικό αυτό πρόβλημα. Ε, ευχαριστώ και θα έχω τη δυνατότητα στην συνέχεια για να προσφέρω και άλλες πιθανές πληροφορίες αλλά και προβληματισμούς που θα συμβάλλουν στο να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο την ευκαιρία που έχουμε. Thank ε, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Τώρα, ένα θέμα επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή Ζούμε μια ιστορική περίοδο. Γιατί. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε αναλάβει νέες αρμοδιότητες, ε, μετα... χάρη στις συνθήκες Λισαβόνας, για πρώτη φορά μπορούμε και εμείς κάτι να πούμε σε αυτό το τομέα. Μέχρι τώρα ήμασταν σαν τη σταχτομπούτα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει όμως και η συγκυρία. Η Ευρώπη γνωρίζει μεγάλη ύφεση άνευ προηγουμένου και η Επιτροπή το θέλει άλλωστε και το πρόγραμμα της Επιτροπής Μπαρόζο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή λοιπόν θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι μία από τις ένας από τους τομείς που μπορούν να δώσουν όθηση στην οικονομία. Εναπόκειται λοιπόν σε εμά να αποφασίσουμε, να υποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία ή απλά και μόνον θα καταδείξουμε ποιες είναι οι δραστηριότητες. Βεβαίω ο προγραμματισμός είναι σημαντικός αλλά χρειάζονται και πόροι. Συνεπώς, πρέπει να προσελκύσουμε οικονομικούς πόρους με βάση ένα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε. Και εδώ θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, τα όσα λέμε θα έχουν σημασία εάν ο τουρισμός δεν είναι μόνο ένας τομέας, αλλά αν γίνει σύστημα. Τότε ο τουρισμός θα βρεθεί στο επίκεντρο πολλών δραστηριοτήτων με θέματα πολιτιστικά, βιοτεχνικά, μεταφορές, τονίζοντα τονίζοντας ε, το φυσικό καλό των χωρών. Αυτά είναι τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Είναι ανανεώσιμοι πόροι που σέβονται το περιβάλλον, το κλίμα, την προστασία των στοιχείων μας. Ο τουρισμός λοιπόν... Ο τουρισμός λοιπόν είναι πολύ σημαντικός όπως είπε ο Σπύρος. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την προσφορά μας. Να υπάρχει μια ειδική προσφορά ώστε να μην υπάρχει μαζική προσφορά διότι τότε τα πάντα είναι κοινά. Πρέπει να επιμείνουμε στον ιδιόμορφο χαρακτήρα του χώρου μας, της παραγωγής μας. Θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, μια τουριστική βιοπικιλότητα. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα διαγωνισμό ιδεών, ώστε να βρεθεί ε, μια διατύπωση αυτών των ενιών. Να τις εκφράσουμε αυτές τις έννοιες και πρέπει να τονίσουμε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, οι πολιτικές ε, κατά τον τραστ, αντιτραστ και η έννοια της αναβάθμισης της πικιλότητες Τρίτον, πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να συνοδεύονται από οικονομικά μέσα, χρηματοοικονομικά μέσα. Τότε θα μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά. Ευχαριστώ πολύ για τους ε, πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Φιντάνσα και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους για αυτά που είπαν. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη έχει τεράστιο δυναμικό στον τομέα του τουρισμού, αλλά δεν υπάρχει ε, συνεργασία διεθνή, διεθνής και διαπεριφερειακή. Μία λοιπόν από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να γίνει μια ανάλυση της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η ευρωπαϊκή συνεργασία. Πρέπει να το επιτύχουμε, ξέρω ότι δεν είναι απλό, το είπαν και οι συνάδελφοι. Ο τουρισμός ούτως ή άλλως συνδέεται άμεσα ή έμεσα με διάφορους τομείς, με διάφορες πολιτικές, επομένως ο συντονισμό είναι αναγκαίος. Συμφωνώ όμως με αυτό που προτείνει και η Κομισιόν. Βεβαίως πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν και πολλές βελτιώσεις. Δεν νομίζω ότι έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δούμε και το θέμα της καινοτομία. Υπάρχουν κάποια σημεία που θα ήθελα να θίξω. Για παράδειγμα, όταν μιλούμε για την ορατότητα, η Κομισιόν μιλά για, την Ευρωπαϊκή, ε, για το Ευρωπαϊκό Σήμα Ποιότητας. Ε, καταρχάς όμως πρέπει να δούμε αν όντως προσφέρει κάποια προσθέμενη αξία μια τέτοια επισήμανση. Γιατί ήδη υπάρχουν διάφορες ε, ταμπέλες, διάφορα σήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ε, σήμα το οικολογικό, άλλα, οπότε ίσως καλό θα ήταν να συντονιστούμε. Δεύτερον, ανταγωνισμός. Η επαγγελματικότητα και η κατάρτιση είναι σαφώς απαραίτητα. Θα μπορούσαμε όμως να ζητήσουμε τη συμβολή και της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης. Η βιωσιμότητα επίσης είναι σημαντική πτυχή. Θα πρέπει να υπάρξει ένας σύνδεσμος με μοντέλα μεταφορών φιλικά προς το περιβάλλον. Και επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας και την πολιτιστική κληρονομιά και να τις ε, δώσουμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Επίσης, οι ηλικιωμένοι πολίτες, άνθρωποι που είναι πάνω από 55, ή αυτοί που έχουν περιορισμένη κινητικότητα, πρέπει να έχουν εύκολη, εύκολη πρόσβαση στα ξενοδοχεία κτλ. Στα πλαίσια του ICT και του ίντερνετ η πληροφόρηση είναι εύκολο να γίνει, οπότε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε τη σχετική οδηγία. Έχουμε μιλήσει πολύ για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Η εμπειρογνωμοσύνη όμως είναι απαραίτητη και ως ε, μέλος της ε, αντιπροσωπείας Euromed θα ήταν σημαντικό να πω ότι πρέπει να δούμε και τις σχέσεις μας με τις μεσογειακές χώρες και πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας ε, επαναλάβω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μιλά για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν χώρες όμορες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να το δούμε. Σίγουρα οι σκιώδεις συγητές ε, θα ε, βοηθήσουν ε, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει στον τομέα του τουρισμού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ράνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, γνωρίζω την ευθύνη που έχω ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και σήμερα μπορώ να πω ότι η... έχει αλλάξει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για την Επιτροπή ε, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Φυσικά το, το θέμα ε, βασίζεται στη δική μας την Επιτροπή στην συζήτηση που γίνεται για, την... για τον εκπαιδευτικό τουρισμό και συζητούμε το πώς γίνεται να συνδέσουμε χώρες μεταξύ τους μέσω του ε, εκπαιδευτικού τουρισμού ή ε, μέσω μαθημάτων γλωσσών ή μέσω άλλων ε, οδών. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με αυτή τη δυνατότητα. Θα μπορούσαμε ίσως να βρούμε λοιπόν κάποιες συνδέσεις και βεβαίως αυτό θα έπρεπε να μπορεί να το χρηματοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα από τα σημεία. Επίσης, μεγάλη αξία έχει και η παιδεία, η εκπαίδευση, το διητό σύστημα συγγνώμη, ε, θεωρίας και πράξης. Ε, μελετά κανείς, σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα γυμνάσιο και έχει τη δυνατότητα, και είναι σημαντικό αυτό, να μπορεί να ταξιδέψει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και σε τρίτες χώρες ώστε να μάθει γλώσσες ε, για να έχει μια ποιοτική ε, εκπαίδευση και να μπορεί να παρέχει στο μέλλον ποιοτικέ υπηρεσίες. Επίσης, Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, το έχουμε κάνει και με άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού, να είναι πιο εύκολος ο τουρισμός, ε, να μην περιμένουμε δηλαδή τους τουρίστες μόνο όταν ε, λάμπει ο ήλιος, ε, να, να προωθήσουμε και το χειμερινό τουρισμό, να δώσουμε ευκαιρίες στους πολίτες. Κάτι που νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο εύκολο αποδεκτό από τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, ο κοινωνικός τουρισμός σε μένα δεν μου αρέσει ως όρος. Θα πρέπει να υπάρχει τουρισμός για όλους, για μεγάλους, για μικρούς, για νέους, για ηλικιωμένους, για όλους. Ε, ακόμη και σε περιόδους ε, οικονομικής κρίσης όπως αυτή που περνούμε τώρα, ε, δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να, να χρηματοδοτήσει νέα προγράμματα τουρισμού. Θα μπορούσε όμως να υποστηρίξει τα υπάρχοντα. Θα μπορούσε να βασιστεί στις υπάρχουσες πλατφόρμες θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε, θα μπορούσαμε να τις γνωστοποιήσουμε περισσότερο και θα έπρεπε. Και βεβαίως στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού είδαμε ότι και ο αθλητισμός είναι ένα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός τομέας. Το, ο αθλητισμός αναγκάζει ουσιαστικά τους ε, ανθρώπους να ταξιδεύουν, οπότε μπορούμε να προωθήσουμε και τον και τον, και τον, ε, και τον αθλητισμό ως κομμάτι του, του τουρισμού. Θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Έχω συζητήσει και με τον ε, συνάδελφο Φιντάνσα και ελπίζω να βρούμε μια κοινή άγουσα μεταξύ των δύο επιτροπών. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι ε, το θέμα αυτό και η Αυστρία πρέπει να πω είναι ότι έχει, είναι η μόνη χώρα η Αυστρία η οποία έχει δύο ε, ε, περιόδους υψηλού τουρισμού και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Οπότε προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία για να μπορέσουμε να πείσουμε περισσότερο και τους πολίτες μας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε μεταξύ των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Φιντάνσα. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το πλαίσιο δράσεων της Κομισιόν θα ήθελα επίσης να το χαιρετήσω. Ούτως ή άλλως ε, είμαστε στην ε, αρχή της ε, επικουρικότητας και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο έχει λάβει αυτή τη νέα αρμοδιότητα για τον ε, τουρισμό. Τα επόμενα χρόνια θα είναι όντως μεγάλη πρόκληση για μας, γιατί προκύπτουν πολλοί νέοι τομείς που θα χρειάζονται αντιμετώπιση και διαχείριση. Ο τουρισμός ούτως ή άλλως είναι διασυνοριακό αγαθό και νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και στην Ευρώπη πολύ περισσότερα διεθνή γεγονότα, οργανισμούς που οργανώνουν διεθνείς αθλητικές ας πούμε, δραστηριότητες, να τις φέρουμε περισσότερο στην, προς την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αν ρυθμίσουμε πάρα πολύ τις ε, τουριστικές ροέ κινδυνεύουμε να εμπλακούμε στα χωράφια της, του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας. Ε, μεγάλες πόλεις, ας πούμε, όπως Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, δεν έχουν πρόβλημα να προσελκύσουν ε, τουρίστες, αλλά ο περιφερειακός τουρισμός πάσχει. Πρέπει να τον προωθήσουμε. Επίσης, τα δικαιώματα των ε, ε, επιβατών είναι πολύ σημαντικά. Όλα αυτά είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να τα διαφημίσουμε ε, από την πλευρά της Ευρώπης. Η παράταση τώρα την, της σεζόν, αυτό ίσως θα πρέπει να γίνει ε, αναομάδες. Ας πούμε θα μπορούσαμε ίσως να συντονίσουμε τις σχολικές ε, διακοπές των ε, σχολείων. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλή πρόταση. Νομίζω ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αν ας πούμε έκαναν διακοπές στα σχολεία και οι μαθητές πηγαίναν μόνο διακοπές στην Γερμανία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. <coughs> Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ. Μιλούμε για τον ευρωπαϊκό τουρισμό και δικαίως μιλούμε, αλλά έχουμε προβλήματα διασυνοριακά. Οι πολίτες ε, παραπονούνται ότι μεταξύ του βαβαρικού δάσους και του ε, τσεχικού και των τσεχικών συνόρων κλείνουν τα περάσματα και δεν μπορεί κανείς να περάσει και να θαυμάσει το δάσος. Θέλουμε να συνδέσουμε την Ευρώπη. Μιλούμε και για τις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Ξέρουμε ότι τα τρένα περνούν τα σύνορα. Πριν από τρία χρόνια είχαμε ήδη αποφασίσει ότι θα έχουμε ένα πρόγραμμα ενημερωτικό για όλες τις υδροδρομικές συνδέσεις, ευρωπαϊκό, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει ένα ε, εισιτήριο, ε, το έχουμε για τις αεροπορικές μεταφορές, ε, θέλαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και με τις σιδηροδρομικές. Δεν έχει γίνει αυτό, γιατί οι ε, σιδηρόδρομοι δεν ήθελαν να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό μέσω ενό ηλεκτρονικού υπολογιστή θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό. Επίσης, ε, είχαμε πει για του επιβάτες, για τα δικαιώματα των επιβατών. Εγώ ε, πάω πολύ συχνά βόλτα με το ποδήλατό μου και αυτός ο τομέας ε, θα μπορούσε να είναι σημαντικός. Ε, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το ποδήλατό του έχει αυξηθεί κατά 20%. Κάποτε έβλεπα πολλούς ανθρώπους με τα αυτοκίνητά τους να πηγαίνουν και τώρα τους βλέπουμε ένα ποδήλατο. Όλους κατά μήκος διαφόρων ποταμών να απολαμβάνουν την βόλτα τους. Ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να προωθήσουμε την... Ε, ε, το, ότι να, το μπορούν οι πολίτε να χρησιμοποιούν και το ποδήλατό του και να το παίρνουν μαζί και στα μέσα μαζικής μεταφορά. Στη Γαλλία πούμε αυτό συμβαίνει. Σε όλα τα, όλα τα τρένα μπορεί κανεί να πάρει μαζί και το, α, και το ποδήλατό του. Και μάλιστα και στα τρένα υψηλή ταχύτητα, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να μπορεί να γίνεται αυτό. Σε κάποια κρατημέλη ήδη γίνεται. Σε κάποια άλλη όχι βέβαια. Στο Eurostar, στο TGV, στο Θαλή μπορούμε να, το, να πάρουμε μαζί το, το ποδήλατο. Δυστυχώ στα γερμανικά τρένα ακόμη δεν έχει γίνει αυτό. Ε, αν θέλουμε λοιπόν ένα βιώσιμο πολιτι... ε, τουρισμό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ε, που έχουμε. Επίσης, χαιρετίζω το ότι ο επίτροπο Τουρισμού έχει δημιουργήσει τους κανόνες για τον, ε, για τον τουρισμό. Υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν τα, τα ποδήλατά τους, πάνε βόλτα στους ποταμούς και τις ε, θάλασσες. Τα Πυρηναία στέκονται βεβαίως ανάμεσα στο δρόμο που, το γνωστό που υπάρχει ε, από, την, ε, από την Ορβηγία ως το Σαντιάγο Δε Κομποστέλα στην Ισπανία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να γίνουν πολλές συνδέσεις. Μπορούμε να συνδέσουμε και τις μεταφορές, την ιστορία, τον πολιτισμό. Όλα αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε και θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, για τις ε, προθεσμίες ε, είναι λίγο με εκπλήσει, γιατί εμείς έχουμε 16 ομοσπονδιακές, ε, ομοσπονδιακά κρατήδια και όλοι, όλα έχουν τελείως διαφορετικές διακοπές. το να κάνουν τώρα όλα τα σχολεία τρεις, τρεις μήνες διακοπές δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Αυτό δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι όταν έχουμε ολομέλεια στην, στο Στρασβούργο, ε, τα, τα ξενοδοχεία είναι δύο φορές τόσο ακριβά. Για, άλλους πάλι, για άλλες, σε άλλες περιόδους πάλι είναι άδεια τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτό που είπε πριν ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα φώτα που μας έδωσε. Πράγματι, όπως υπόθηκε, ο τουρισμός είναι μία δραστηριότητα που αντιστάθηκε στην κρίση και έχει, παρουσιάζει ακόμα ευκαιρίες. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας πάνω σε ένα σημείο. Έρχομαι από το Μομπλό και αυτή η περιοχή πηγαίνει μέχρι τη Μεσόγειο και λόγω της αλλαγής των κλιματικών συνθήκων ε, είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Σε ορισμένες περιοχές βλέπουμε τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών και πιθανό να υπάρξουν ε, προβλήματα με την κατάσταση της ε, τουριστικής δραστηριότητα σε δύο ε, κλίμακα τα προσεχέτη. Με ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίω έχουμε είναι πώ να διατηρήσουμε την τουριστική ποιότητα. Και υπογραμμίζω τη σημασία που έχει η εκπαίδευση του προσωπικού και ακόμα και η τυποποίηση, αν θέλετε, παρόλο που θα πρέπει να υπάρχει επικουρικότητα των χωρών, σημαντικό είναι να έχουμε απέναντι στον, στους τουρίστες όλου του κόσμου ε, μια χάρτα ποιότητας που θα είναι τυποποιημένη για όλους τους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Ευχαριστώ. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, deviza Uniți în diversitate caracterizează Europa. Ευχαριστώ. Εμείς εδώ έχουμε ένα ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Και όποιος έρθει στην Ευρώπη ε, βλέπει ότι υπάρχει μια πολιτική ποικιλότητα και ε, ότι μπορεί κανείς εύκολα να ταξιδέψει από τη μία πρωτεύουσα στην άλλη και μεταξύ των πόλεων και ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλότητα πολιτιστικής μορφής σε έναν μικρό χώρο. Ο πολιτισμός, η κουλτούρα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης. Πιστεύουμε, συνεπώς, ότι όλο και περισσότερο θα πρέπει να συνδέσουμε ε, τα εθνικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. τώρα ως προς την προστασία των καταναλωτών, θα ήθελα να πω το εξή ε, στην Επιτροπή και να τη ρωτήσω πότε ε, θα προετοιμάσει ένα πακέτο τουρισμού. Γνωρίζουμε ότι ε, στη Σόλβιτ πολλά παράπονα, αν θέλετε, αφορούν τον τουρισμό. Εάν λοιπόν θέλουμε να αναπτύξουμε τον ευρωπαϊκό τουρισμό, πρέπει να βελτιωθούν και οι τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται. Κύριε Πρόεδρε, όταν ε, η αντιπροπία μας μετέβη στη Μαγιόρκα, επισκεφθήκαμε μια ανώτερη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ε, μιλήσατε για το πρόγραμμα Καλυψό και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν και εθνικά προγράμματα παράλληλα με τα κοινοτικά προγράμματα. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχουμε λάβει αρκετά υπόψη μας. Τον ε, τουρισμό, γιατρικ... Ε, γιατρικής μορφής, τα σπα. Διότι νομίζω ότι αυτά τα σπα θα μπορούν να αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, ευχαριστώντας τον συντονιστή. Πρόκειται για ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι ε, μεγάλο το βήμα, αλλά νομίζω ότι θα αποδώσει αυτή η επιτροπή ε, δεν θα έπρεπε να ονομάζεται Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών, διότι όπως είπαμε ο τουρισμός είναι σταχτομπούτα. Και ε, στο παρελθόν, όταν είχαμε και την περιφερειακή ανάπτυξη, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ο επιχειακός χαρακτήρας του τουρισμού αναφέρθηκε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ισχυρά μας σημεία, διότι το χειμώνα υπάρχουν πολλές επιλογές. Μιλήσατε για την, τις πολλές δυνατότητες επιλογής, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θέλει ο καταναλωτής. Ορισμένοι καταναλωτές θέλουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας, άλλα θα θέλουν τα ξενοδοχεία δύο ή τριών αστέρων, άλλοι πάλι θα θέλουν τα πανδοχεία, ε, το bed and breakfast. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο, αν θέλει να πάει για κάμπινγκ, να έχει καλές εγκαταστάσεις κάμπινγκ, να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες. Το δεύτερο αφορά την ποικιλότητα και τις επιλογές. Όσον αφορά ε, διάφορους όπως το γκολφ. Ορισμένοι πηγαίνουν στο γκολφ το οποίο είναι φθηνό σε ορισμένες χώρες και πολύ ακριβώς σε άλλες. Ας πούμε, ε, ε εμείς έχουμε εννέα γκολφ σε μια πολύ μικρή, μικρή έκταση. Τώρα πάλι ε, πρέπει να δείτε Τώρα, γιατί τα, στοιχεία. Νομίζω ότι τα πολιτιστικά στοιχεία είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν 27 χώρες οι οποίες έχουν διάφορους πολιτισμούς και θα πρέπει να τονίσουμε την ποικιλότητα μέσα στην ενότητα. Βεβαίω, έχουμε ένα μοσαϊκό πολιτισμών. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Τώρα, η εποχικότητα και πολλοί πηγαίνουν το χειμώνα επειδή βρίσκουν ε, χώρους όπου μπορούν να περπατήσουν και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα συνδυάσουμε. Αποφασιστική σημασία όμω είναι σε εποχή οικονομική κρίσης να είμαστε ανταγωνιστικοί ως προ τις τιμές μας και νομίζω ότι αυτό έχει ε, αντιμετωπιστεί όσον αφορά τι αεροπορικές μεταφορές όπου υπάρχει μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά θα πρέπει να δούμε και στου άλλου τομεί τι θα γίνει. Α πούμε η Ryanair, οποιοδήποτε, ε, οποιαδήποτε εταιρεία είναι ανταγωνιστικέ. Εδώ έχουμε καλές τιμές. Ε, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην αγορά και ω αποτέλεσμα τη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα έχουμε πρέπει να έχουμε μείωση των τιμών. Ένα από του τομεί, τους οποίου θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τις νέες αγορές. Η περιοχή μου λέγεται ότι πάρα πολλά, ε, άτομα στι ΗΠΑ ε, ε, είναι Ιρλανδική καταγωγή. Λοιπόν, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την αγορά στι ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί θέλουν να βρουν τι ρίζε του, από πού προήλθαν, θέλουν να επιστρέψουν στη γη του. Γι' αυτό α πάρουμε τον Ομπάμα ω παράδειγμα, ο οποίο έχει και εκείνο Ιρλανδικέ καταβολέ. Γι' αυτό αξιοποιήσαμε πολύ καλά αυτή την αγορά. Εκεί όμως που σκοτώσαμε την με τα χρυσά αυγά ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλη, υψηλές οι τιμές μας. Είμαστε πολύ ακριβοί. Έχουμε ένα καλό προϊόν, αλλά δεν πρέπει να είναι πολύ ακριβό. Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχουν λιγότεροι περιορισμοί για τις βίζες. Ήταν πολύ σωστό αυτό που υπόθηκε. Θα μπορούσαμε να έχουμε αμοιβαία ανταλλαγή σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν 20 εκατομμύρια ε, στην Ταϊουάν που ε, μπορούσαν να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά τώρα με του περιορισμού που υπάρχουν ε, δεν θα έρχονται. Γι' αυτό πρέπει να δούμε το θέμα τη βίζα. Καλά ξεκινήσαμε. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Αλλά θα βγουν πολλά καλά σε περίοδο οικονομική κρίση ιδίω. Ευχαριστώ. Thank you. Before I bring in the uh, commission... πριν, πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φιντάνσα για να κλείσει. Ήταν πολύ καλή η εισαγωγική σας παρουσίαση. Θα ήθελα όμως να κάνω και τρεις παρατηρήσεις. Καταρχήν πρέπει να διευρύνουμε τον τουρισμό μας για να συμπεριλαμβάνει και άλλα είδη πέρα αυτών των παραδοσιακών, δηλαδή βουνά το χειμώνα και παραλία το καλοκαίρι, να αλλάξουμε φιλοσοφία. Και σχετίζεται αυτό με κάτι που είπε και η κυρία Ράνερ για την Επιτροπή Πολιτισμού που συζητά το θέμα της βιομηχανικής παράδοσης, της πολιτιστικής παράδοσης, τον αθλητικό τουρισμό. Εγώ όταν ε, φεύγω τη Δευτέρα από το Μάντσεστερ, κάνω, στην ουρά βλέπω πολλούς Δανούς, Σουηδούς, Νορβηγούς, που έχουν έρθει στην Αγγλία για να δουν τη Λίβερπουλ να παίζει ή την Everton ή τη Manchester City και γυρίζουν στην πατρίδα τους. Οι Δανείοι και οι... Ε, ξέρεις, δεν είναι εποχή του ράγκμπι τώρα, για ποδόσφαιρα έρχονται. Είναι ε, συγκλονιστικό όμως το πόσος κόσμος έρχεται για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδας του. Υποθέτω ότι δεν είναι το επίπεδο των των, του αθλητισμού σε αυτές τις χώρες εξίσου υψηλό όσο το Premier League, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δεύτερον, αυτή η οδηγία για τα πακέτα διακοπών έχει, είναι πλέον παροχημένη. Έχει ξεπεραστεί τελείως. Και μάλιστα στρεβλώνει και τον ανταγωνισμό σε μερικές περιπτώσεις. Γιατί οι tour operators, οι TUI, ο Thomas Cook, ε, η Thompson δεσμεύονται από αυτή την οδηγία, αλλά η Ryanair δεν δεσμεύεται. Θα σας πουλούσαν βεβαίως ένα πακέτο διακοπών στην ιστοσελίδα τους, ε, πουλώντας σας βεβαίως μεμονωμένα τα διάφορα τμήματα του πακέτου. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι η ώρα να ε, καταλήξουμε σε μια νέα οδηγία που θα συμπεριλαμβάνει και τα δικαιώματα των επιβατών, όπως είπα και διάφοροι συνάδελφοι. Τρίτον, δεν υπάρχουν ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφάλειας στα διάφορα ξενοδοχεία και διάφορες εγκαταστάσεις στέγασης στην Ευρώπη. Έχουμε ορίσει ελάχιστα, ελάχιστους ε, όρους ε, πτήσεων για τα πληρώματα των ε, αεροπλάνων, ελάχιστες ώρες οδήγησης για τους, για τους οδηγούς φορτηγών, ελάχιστα πρότυπα για τα οχήματα. Δεν έχουμε ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας για τα ξενοδοχεία στην Ευρώπη. Και αν δείτε και τα δυστυχήματα που συμβαίνουν, Δύο παιδιά ε, σκοτώθηκαν, ας πούμε, στην, ε, στην ε, Κέρκυρα από δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. σε, ένα, σε ένα μεγάλο παρεσινό ε, ε, ξενοδοχείο πιασε φωτιά. 18 άνθρωποι επίσης πέθαναν και 20 τραυματίστηκαν. Στα, στη Κανάρια επίσης πνίγηκαν σε μια πισίνα τουρίστες. Όλα αυτά τα έχουμε δει. Το 2008, κύριε Φιντάντζα, η Επίτροπος Κούνεβα εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Ξενοδοχείων, τον κλάδο των ξενοδοχείων, να ε, ορίσει τέτοιο, τέτοια πρότυπα για την ασφάλεια, έχοντας ε, την πρόθεση αυτά να υπογραφούν από τους ξενοδόχους. Ε, το τέλος του 2009 αποφάσισαν ότι θα, ε, δεν θα προχωρήσει η χάρτα αυτή, κάνοντας την απολύτω ε, επιφανειακή, απολύτω άχρηστη. Τώρα λοιπόν δεν έχουμε καμία χάρτα, δεν έχουμε τίποτα νομικό δεσμευτικό, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μα. Οπότε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα έχουν ε, ε, αποτύχει απόλυτα. Δείτε το λοιπόν και αυτό στα πλαίσια της έκθεσης σας. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Τουντίνη είναι εδώ, νομίζω. Ναι, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια για να σας ευχαριστήσω την πρόσκλησή σας να παρακολουθήσω αυτην την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ευχαριστώ και τον κύριο Φιντάντσα για την ε, ενδιαφέρουσα πρόταση την οποία Σημεριζόμαστε τον αφορά την δομή, της προτεραιότητες και θα ήθελα να προσθέσω ότι θεωρούμε ότι η ανακοίνωσή μας είναι πάρα πολύ φιλόδοξη, πάρα πολύ περιεκτική, αλλά σήμερα είδαμε ότι παρασιάζονται πολλές ιδέες καινούργιες. Άρα υπάρχει ε, περιθώριο να συμπεριλάβουμε στην πρότασή μας και νέες ιδέες. Περιμένουμε λοιπόν την έκθεση ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε το σχέδιο εφαρμογής το οποίο βρίσκεται σε επεξεργασία και σήμερα εφόσον είμαι εδώ Ήδη έχω καταγράψει κάποιες από τις ιδέες οι οποίες εκφράστηκαν για να τις λάβω υπόψη. Σε σχέση τώρα με το θέμα της αναδεώρησης της οδηγίας για το πακέτο υπηρεσιών το τουριστικό, σε ένα χρόνο θα έχουμε τη νέα πρόταση του χρόνου Δηλαδή το Σεπτέμβριο, δηλαδή του 2011. Ευχαριστώ κύριε Σουντάντση, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις πολύ θετικέ τους παρατηρήσεις και για τη συνεισφορά τους. Και βεβαίως όπως σας είπα, σε πρώτη φάση θα προσπαθήσω στις επόμενες εβδομάδες να συγκεράσω όλες αυτές τις ιδέες για να παρουσιάσω ένα γραπτό έγγραφο το οποίο θα μελετήσουμε εκ των ιδέων. Άκουσα πολλές ιδέες από όλους τους ε, συναδέλφους και πρέπει να πω ότι όλα αυτά με ενθαρρύνουν στο να εντείνω τις προσπάθειές μου για να εκπονήσω την έκθεσή μου. Προηγουμένως είπα τι έχουν κάνει για τα άλλα θεσμικά όργανα, αλλά ξέχασα να αναφέρω τη Βελγική Προεδρία, συγγνώμη, η οποία θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι μία από τις προτεραιότητές της. Επίσης, ξέρω ότι η επόμενη Προεδρία, η Ουγγρική, θέλει επίσης να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση και θεωρεί τον τουρισμό ως ένα τομέα δράσεων προτεραιότητας. Όπως είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι για μας Αυτό το οποίο είναι σημαντικό δεν είναι να κάνουμε μία έκθεση στην οποία θα παριθμίσουμε τα είδη του τουρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει, το έχουν, έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό διάφοροι συνάδελφοι στο παρελθόν. Αυτό το οποίο θέλω εγώ να κάνω είναι μαζί με τους άλλους συναδέλφους να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις ώστε να αναπτυχθούν όλοι οι τουριστικοί τομείς και διάφορες μορφές τουρισμού και να μπορέσουμε να έχουμε μια κάποια πρόοδο σε σχέση με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα τώρα να πω το εξή στους συναδέλφους που ανέφεραν το θέμα της επικουρικότητας. Στην συνθήκη της Λισαβόνας είναι απολύτω αυτή τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ε, διευκρινήσεις σχέση με αυτό το θέμα, παρά το γεγονός ότι ακόμη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο υπάρχει αρμοδιότητα για θέματα τουρισμού. Βεβαίως μπορούμε να λάβουμε υπόψη την αρχή αυτή, όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Και τώρα θα ήθελα να κάνω κάποια ε, σχόλια. Το θέμα της κατάρτισης, της επιμόρφωσης είναι σημαντικό. Θέλουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό άλμα. Δεν θέλουμε να υπάρχει μόνο για τους σερβιτόρους, για τις σερβιτόρες η σωστή κατάρτιση. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε και σωστούς επαγγελματίες ε, σε αυτούς που αφορούνται με διαχείριση, διαχείριση των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τον τουρισμό. όσον αφορά το θέμα των συνεργειών. Είπαμε. Κάτι για τα πακέτα, τα all inclusive. Και είπα ότι θα πρέπει εμείς να υποφεληθούμε από την πρόοδο της τεχνολογίας, διότι το ίντερνετ είναι ένα μέσον το οποίο χρησιμοποιούν όχι μόνο ο καθένας από εμά που είναι τουρίστας, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προβάλλουν τα προϊόντα τους και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το ίντερνετ και για αυτές. Όσον αφορά τις βίζα, τις θεωρήσεις, έχουμε δυνατότητες πάρα πολλές, διότι έχουμε δυνητικούς τουρίστες από πολλές χώρες, Φερρυπίν, από την Κίνα ή από την Ρωσία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να επισκεφθούν, να γνωρίσουν την Ευρώπη. Και η ιδέα ε, προώθησης της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού είναι μια εξαιρετική ιδέα. Βεβαίως, πάντα θα υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης και των πόλεων της Ευρώπης, αλλά η βασική επιλογή σε πρώτη φάση για τον Κινέζο θα είναι πού επιλέγω να πάω, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην ε, Αφρική, Φερρυπίν. Όπως είπε και η εκπρόσωπος της ε, ε, Εκτελεστικής Επιτροπής, η θα γίνει του χρόνου η θεώρηση τη ε, οδηγία για τα πακέτα, τα all inclusive, αλλά αυτό το οποίο είναι παράξενο είναι ότι δεν θα είναι υπεύθυνο πλέον ο κύριο Ταγιάννη, που είναι υπεύθυνο τον τουρισμό, αλλά η κυρία Ρέντινγκ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι δραστηριότητε, οι τουριστικέ, αφορούν πολλού επιτρόπου, κατακαιρματίζονται κατά κάποιο τρόπο. Και ίσως αυτό δυσχεραίνει κάπως τα πράγματα, διότι έχουμε απέναντί μας διαφορετικούς ε, συνομιλητές και πολλές φορές είναι δύσκολο όταν υπάρχουν διάφοροι ε, συνομιλητές να παρεύουμε εύκολα. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε το συντομότερο δυνατό. Θα σας υποβάλω την εκθεσή μου. Σας ευχαριστούμε. Περιμένω να παρουσιάσετε το σχέδιο εκθεσή τον Ιανουάριο. In... Κατόπιν θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή το Μάρτιο και κατόπιν στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση του κ. Φεντάντζε. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα μας τώρα στην ημερήσια διάταξη είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 2007-2013. Ο κ. Σκόλετζεκ σας σχέδιο γνωμοδότησης. Δεδομένου ότι ο κ. Τζέκ δεν είναι εδώ. Η κυρία Βίλσον αντικαθιστά, αλλά και εκείνη είναι απούσα. Συνεπώς, εναπόκειται στον Πρόεδρο να παρουσιάσει επισήμως τη γνωμοδότηση την οποία έχετε στο φάκελό σας, αριθμός 4. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την go into the... σχέδιο γνωμοδότησης πρωτού αρχίσει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, γνωρίζετε ο κ. Σκόλατσεκ, προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με την γνωμοδότηση την οποία έχω εγώ υποβάλει για την Επιτροπή ε, σχετικά You will note from... σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα ο κ. Κόλετσέκ υπογραμμίζει το 82 δισεκατομμύρια ευρώ των ε, διαθροτικών ταμείων ε, θα διατεθούν το 2007-2013 για τις μεταφορές, τα μισά όμως για τα προγράμματα TEN-T, 17 δισεκατομμύρια για τα δίκτυα προτεραιότητας TEN-T και 27,2 δισεκατομμύρια για το άλλο μέρος. Τα άλλα μισά θα επενδυθούν σε περιφερειακά τοπικά προγράμματα, όχι ε, για το TEN-T. Επίσης, ε, υπενθυμίζω ότι δεν υπάρχει ισορροπία ε, όσον αφορά τις επενδύσεις μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς και αναφέρεται στην καθυστέρηση αυτών των διασυνοριακών προγραμμάτων και τελικά πιθανόν το πρόγραμμα TEN-T θα περιέχει απλά 27 εθνικά δίκτυα. Ε, τα αγγλικά του κύριου Κόρσουκ φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μου αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Επίσης λυπούμεθα, διότι όταν ε, στα πλαίσια του προγράμματος συνοχής ε, η ανισορροπία η οποία υπάρχει μεταξύ των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών θα συνεχιστούν αν καθυστερήσουν οι επενδύσεις στο δίκτυο, όπως αναφέρεται ε, στο, ε, στην έκθεση του 2010. Και αν δούμε ε, ότι υπάρχει μια προκατάληψη κατά των οδικών μεταφορών επίσης, ανησυχεί επειδή δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες όσον αφορά τις επενδύσεις που γίνονται και επίσης ε, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει καλύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής όσον αφορά ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και επίσης υπογραμμίζει ότι με βάση την οικονομική κρίση θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα. Επίσης υπογραμμίζει την ε, προστιθέμενη αξία αυτών των δικτύων κυρίως στα ε, διασυνοριακά τμήματα και στη διασύνδεσή τους με τα προγράμματα σιδηροδρόμων και πλωτών οδών. Επίσης, ε, ζητεί να γίνονται ε, σωστή χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα και να υπάρχει ένα ποσό για τα βασικά δίκτυα ε, των ευρωπαϊκών, ώστε να χρησιμοποιείται αποτελεσματικότερα η χρηματοδότηση ώστε να υπάρχουν στόχοι πιο βιώσιμοι και πιο καλή εφαρμογή του δικτύου. Εξ ονόματος του κυρίου Κάλατσέκα παρουσίασα αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και έχουμε πρώτα τον κύριο Ήταλα. Thank you, I can uh, mainly agree with the rapporteur and uh, very important to emphasize. Μπορώ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον εισηγητή για την πολιτική συνοχή. Ειδικά όταν μιλούμε για τα προγράμματα τα διασυνοριακά. Πρέπει να συζητήσουμε και για τα σύνορα από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο εισηγητής για τις ε, εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις ε, κλιματικές αλλαγές και τις εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, επειδή εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Ελέγχου του Προπολογισμού, είναι ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνουμε όλα τα δεδομένα. Ε, κάποιοι έχουν ένα πολύ μεγάλο περιθώριο λάθος και ούτε καν επιστρέφουν τα χρήματα που λαμβάνουν. Νομίζω ότι θα πρέπει και αυτό να το θίξουμε. Κάτι τελευταίο, Πρόεδρε. Για την συνεργασία θα ήθελα να λέμε ότι ζητούμε μεγαλύτερη συνεργασία με την Επιτροπή Ρέτζι για, την, για τον τομέα των μεταφορών. Ίσως έτσι να μπορούσαμε λίγο να διασυνδέσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Ιταλά, πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο που είπατε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Να έχουμε και επαφές με, ε, τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων. Ο κύριος Αλχαντράου έχει το λόγο. Ε, περιοριστείτε αν θέλετε στα τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Ο κύριος Λιμπεράσκη δεν μπορούσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Εμείς ε, ευχαριστούμε τον συγκεκριτή, συμφωνούμε με την γνωμοδοτησία του, δεν έχουμε ιδιαίτερα σχόλια να κάνουμε. Συμφωνούμε και με αυτό που λέει. πολλά, από τα ταμεία, πολλά κονδύλια από τα ταμεία συνοχής ε, δαπανώνται στις ε, οδικές ε, μεταφορές. Και αν δείτε τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σιδηροδρομικές δεν έχουν αρχίσει καν και για τα συνοριακά προγράμματα και για τις ε, παραμεθόριες περιοχές, ε, αυτό είναι πρόβλημα και θα πρέπει να το τονίσουμε. Θα ήθελα επίση να αναφέρω μια τροπολογία του συναδέλφου για το χαμηλό επίπεδο πληρωμών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Είμαστε περίπου στα μισά της ε, περίοδου από το 2007 και έπειτα. Και βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, το ποσοστό που έχει ε, προβλεφθεί. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Λίφτεμπεργκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας αναφέρω και εγώ ότι συμφωνώ με τις ιδέες του κυρίου Κόλατσεκ, ειδικά με το σημείο 6. Ε, το ζητούμε εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει ε, μία καταγραφή, μία ενίσχυση ε, των ε, ε, τις σχέσεις που υπάρχει μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο, μέχρι στιγμή δεν το έχουμε. Να κάνουμε μια λεπτομερή ανάλυση για το πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να επηρεάσει τον τομέα αυτό. Και όχι μόνο για τι ε, ε, λεπτομέρειες, αλλά και για, το, για, το συνολικό, για τα συνολικά κονδύλια που πάνε στις, στις μεταφορές. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό αυτό. Εδώ χρειαζόμαστε συντονισμένες πληροφορίες, ώστε να, είμαστε, να είναι σαφή τα πράγματα για το τι γίνεται και πώς θα προχωρήσει μέχρι το, το τέλος των, της προγραμματικής περίοδου που έχουμε ορίσει, για, πώς μπορούμε, για να δούμε πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτά που έχουμε οραματιστεί. Με το ερώτημα τώρα των, του, τομείου για τις μεταφορές, ε, ε, δεν είναι Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερη φαν, αλλά ειδικά στις χώρες συνοχής, σε ό,τι αφορά την βελτίωση των υποδομών, θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καθόλου γενική εικόνα, δεν θα μπορούμε καν να ελέγξουμε τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εκεί. Οπότε ε, το είχα πει βέβαια αυτό και στην συζήτηση ε, ήδη που έχει γίνει για το Ταμείο για τις Μεταφορές. Επίσης υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις. Εγώ νομίζω ότι από αυτό που λέει ο συνάδελφος Κόλιτσεκ για τις συνδέσεις ε, των διαφόρων φορέων μεταφορών είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι τα κενά και τα ελλείμματα μεγαλώνουν, αυξάνονται αντί να μειώνονται. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Φλάσο και είναι σκιώδης εσείς; Δεν μπόρεσε όμως να έλθει σήμερα. Γι' αυτό θα κάνω εγώ κάποιες παρατηρήσεις ε, εκ μέρους του. Ο συνάδελφος Φλάσοκ θέλησε να καταθέσει διάφορες τροπολογίες. Όπως λέει στην παράγραφο 3 ο συγγετής, όντως υπάρχει έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των κονδυλίων που χορηγούνται για τα διάφορα είδη μεταφορών διαφορετικά. Θα πρέπει όμως να δούμε ποια είναι η επιλογή την οποία κάνει κάποια χώρα. Δίδεται προτεραιότητα στα εσωδικές μεταφορές αντί στις πλωτές για κάποιον. Σύμφωνα με την παράγραφο 7, επίσης, πιστεύω ότι δεν αναφέρονται οι οδικές μεταφορές, αναφέρονται οι εσωτερικές πλωτές ε, ε, διαδρομές και οι σιδηρόδρομοι, σιδηροδρομικές. Αλλά νομίζω ότι το ενίσχυση του οδικού δικτύου επίσης σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει μια ολόκληρη περιοχή. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι ο κύριος Φλάσιαχ επίσης θα καταθέσει και άλλες τροπολογίες. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα κάνω τέσσερις παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα. Εδώ και κάποιο καιρό ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μεταφορές για την συνοχή και τον Πόσο σημαντική είναι η συνοχή για την ανάπτυξη των μεταφορών, όχι για τους ιδίους λόγους και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναφέρει πολύ σωστά στην εκθέση του κ. Φλασάκ. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Πού είναι τα χρήματα των μεταφορών. Τα χρήματα των μεταφορών βρίσκονται στη Ρέτζιο, όχι στη δική μας Επιτροπή. Διότι φαίνεται ότι εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επηρεάσουμε κατά 1,5% τα ποσά τα οποία μπορούν να επηρεάσουν οι συνάδελφοι της Ρέτζιου. Τρίτο. Όποιος πληρώνει έχει τον πανολόγο. Άρα αφού πληρώνει η Ρέτζιο και είναι υπεύθυνη, εκείνη έχει τον πανολόγο. Αυτό το είπαν διάφοροι συνάδελφοι. Τα είδη μεταφορών τα οποία ε, ευνοούνται ή δεν ευνοούνται, εξαρτώνται από ποιος πληρώνει. Πολλές φορές όχι τα οδικά δίκτυα, πολλές φορές ναι. Τα κριτήρια για την περιφερειακή ανάπτυξη επίσης, άρα η χρηματοδότηση εξαρτάται ποτέ του ίδιους κριτήρια. Και τέταρτη παρατήρηση, τελικά όλοι λένε ότι για να δαπανώνται σωστά και κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα χρήματα τα οποία αφιερώνονται στις μεταφορές πρέπει να τα βρούμε με αυτούς οι οποίοι δίνουν τα χρήματα. Αυτό όμω δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ε, αρέσει κανέναν. Ε, δηλαδή, αν ε, κάποιος σύμφωνα με τους υπεύθυνους του προπολισμού έχει κάποια χρήματα να μοιράσει, δεν θέλει να έρθει κάποιος άλλος να του πει δώστε εδώ ή δώστε εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί. Πρέπει όμως εμείς με διπλωματικό τρόπο να χειριστούμε το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν ήπιο τρόπο συντονισμού με την Ρέτζιο. Επίσης θα πρέπει εκτός από αυτό τον συντονισμό να μπορέσουμε εμείς για την βελτιστοποίηση των μεταφορών να προσθέσουμε κάποια ε, στοιχεία. Κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν ε, την ε, τέχνη που πρέπει να υπάρχει για να γίνονται σωστά οι μεταφορές και να μπορέσουμε να πάρουμε το μέρος μας κατά κάποιο τρόπο και αυτούς οι οποίοι δίνουν τα χρήματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, το ποιος δίνει και πού τα δίνει και με ποιον τρόπο τα δίνει τα χρήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και βεβαίως με συντονισμό επαναλαμβάνω με τους ε, συναδέλφους περιφερειακής ανάπτυξης και ενδεχομένως τους συναδέλφους Επιτροπής Προϋπολογισμών μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρος. Θα είμαι σύντομο Πρόεδρε για την συνοχή και τις μεταφορές. Ξέρουμε ποια είναι η σχέση που υπάρχει 80% οδικές μεταφορές και 20% για τα υπόλοιπα. Τα δεδομένα που έχουμε είναι και προκύπτουν από τα έγγραφα που έχουμε. Για τα ε, διευρωπαϊκά, ε, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μιλούμε για 10 φορές περισσότερα από τα εθνικά δίκτυα, ειδικά για τα, για τα διευρωπαϊκά. Ο όρος λοιπόν που χρησιμοποιεί η Κομισιόν αυτή την όρο της αρεσιμότητας που σημαίνει ότι η, τα κονδύλια θα δίδονται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε ό,τι αφορά αυτές τις προϋποθέσεις νομίζω ότι η συνεργασία και η συνέπεια με την πολιτική α, ε, μεταφορών θα πρέπει να είναι δεδομένη. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε την ε, εντύπωση ότι κάνουμε ένα hold-up, ότι κατακρατούμε τα χρήματα χωρίς να τα δίνουμε. Απλώς θέλουμε να έχουμε περιφερειακή πολιτική, σωστή, ε, περιφερειακή ανάπτυξη και αυτό μπορούμε να το συνδέσουμε και με τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Να γίνεται δηλαδή παράλληλη δουλειά ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και αντιθέσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs.

προσελκύσουμε κεφάλαια προς τις μεταφορές. Η ανάλυση μας κατέδειξε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εμπειρία όσον αφορά ε, τη διάθεση κονδυλίων σαν τα και πρέπει να υπάρξουν τα απαραίτητα κονδύλια για τη διευρωπαϊκά δίκτυα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα είτε τα εθνικά κεφάλαια είτε τα κεφάλαια του Ταμείου Συνοχής. σε αυτή τη γνωδότηση γίνεται προσπάθεια χρησιμοποίηση ε, των πόρων από το Ταμείο συνοχη Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι σε αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να υπογραμμιστεί η συμπληρωματικότητα των πηγών χρηματοδότησης έχουμε ε, τον προπολογισμό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά ε, και τα άλλα κονδύλια. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Για αυτό που είπε ο συνάδελφος Γκρός. Φυσικά μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε και να διαφωνήσουμε. Αλλά όταν έχουμε 80% υποδομές οδικών μεταφορών για το διαφορετικό ε, ταμείο και 20% ε, ε, το Ταμείο για τα Διευρωπαϊκά Διεκτυά, τότε δεν έχουμε κερδίσει τίποτα για το κλίμα. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πού πάνε τα λεφτά. 60% για τις οδικές και τα υπόλοιπα για τους, ε, για τους σιδηροδρόμους εγώ έλεγα. Τώρα βλέπω ότι είναι 80% με 20%. Ευχαριστώ που μου το λέτε. Στο πρώτο πακέτο για τους σιδηροδρόμους είχαμε συμφωνήσει εάν θυμούμε καλώς, ότι τουλάχιστον 40% θα πάει στους σιδηροδρόμους. Και αυτό μπορούμε να το δούμε και στην, ε, το είχαμε πει και στην ε, ψηφοφορία. Εμείς πάντα θέλαμε 40% ε, στην, στους, στους σιδηρόδρομους, 20% στις οδικές μεταφορές και 15% στους πεζούς και στα ποδήλατα. Αν έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο όριο, ανεξάρτητα από το πώ δαπανώνται τα χρήματα και αν έχουμε 40%, αν έχουμε ένα ορισμένο 40%, τότε αυτό, αυτά τα 40% των κορδιλίων θα πηγαίνουν κάπου σωστά. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε όλα στις οδικές μεταφορές. Γιατί ούτως ή άλλως οι περισσότερες ε, ε, εκπομπές αερίων παράγονται από τις οδικές μεταφορές. Αύριο λοιπόν, αν θέλετε, μπορούμε να δείξουμε κατά πόσο θέλουμε να κινηθούμε προς σωστή κατεύθυνση στην ψηφοφορία ή αλλιώ αν θέλουμε να τα αφήσουμε τα πράγματα ω έχουν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Michael. Now, we were at this λοιπόν, δεν βλέπουμε κανέναν από την Επιτροπή στην οποία θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο. Κρίμα, απογοητευτικό, ας πούμε. Γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 8 Δεκεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει το Φεβρουάριο. Συνεπώς, όπως είπαμε, η καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι η 8η Δεκεμβρίου. Το επόμενο θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Αστική Ατζέντα και η Μελλοντική Πολιτική Συνοχής. Η κυρία Ροσμπάχα έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Έρχομαι από την Επιτροπή με την Κορέα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν πολύ καλές τροπολογίες. Πολλά θέματα όμως τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη. Ο κύριος Φεντάλ, μίλησε για τα πλοία ε, στους ποταμούς και επίσης για τα οχήματα στη δική μου την πόλη. Άλλοι μιλήσαν για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Είμαι ευγνώμων για όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ελπίζω ότι βλέπετε ε, πώς θα γίνει η ψηφοφορία αύριο. Υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που θα ήθελα να σας πω. Η κυρία Τίκα με την τροπολογία υπαριθμών 6 ε, ζητάει μια νέα παράγραφο. Συμφωνώ, δεν υπάρχει θέμα. Θα δείτε, όπως είπε ο κ. Κράμερ, Ζήτησαμε ξεχωριστή ψηφοφορία και ζητήσαμε να πάρουμε την τροπολογία του κ. Κράμερ, όχι να την διαγράψουμε από, την, από το συμβασμό, ή ε, αλλά να το, την προσθέσουμε ώστε να υπάρχει το cash sharing και το car δηλαδή ε, να ταξιδεύει κανείς το ίδιο αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Νομίζω ότι τελικά καταλήγουμε σε καλούς συμβιβασμού και όλοι ελπίζω να είναι σε θέση να υποστηρίξουν αυτό το συμβιβασμό μας, διότι αγωνιζόμαστε για αυτούς τους συμβιβασμούς και ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν όλοι και ελπίζω ότι η γνωμοδότηση αύριο θα είναι καλή. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Rike, for the e. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε, η οποία έχει σωστά οριοθετήσει τη συζήτηση. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική, επειδή Φύγει κάτι το οποίο παράδοξα στα ευρωπαϊκά πλαίσια που δεν τολμάει να φτάσει στο κέντρο των πόλεων, ενώ οι πόλη είναι κάτι το πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, εφόσον όμως το 95% ε, του πληθυσμού της Ευρώπης ζει στις πόλεις, αλλά εκεί τα, τα πράγματα δεν συμβαίνουν όπως θα έπρεπε, όπως συμβαίνουν αλλού. Γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον είδαμε το γεγονός ότι οι πολιτικές μετακίνηση στην πόλη, τα προβλήματα συμφορήσεων ε, και τα λοιπά είναι πολύ σημαντικά, διότι ε, το θέμα της μετακίνησης στην πόλη έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία και έχει σχέση με τα δίκτυα προτεραιότητας. Γι' αυτό, αυτό αποτελεί συνέχεια ε, της έκθεσης του κ. Σαβαρίν πριν από λίγο καιρό δεν έχουμε καμία αντίρρηση με την συγκήτρια, συμφωνούμε με τους συμβασμούς που προτείνει και θα τους υποστηρίξουμε. Κατόπιν θα έλεγα ότι υπάρχουν ορισμένες προσθήκες που έγιναν επειδή η έκθεση καθοδηγούσε μεν, αλλά άφηνε ευελιξία ε, για να φύγουν και άλλα θέματα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν συμφωνούμε με το γενικό τόνο της έκθεσης και με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Uh, voorzitter. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και τη κυρία Αγιάλα που δεν ε, μπόρεσε να είναι παρούσα σήμερα. Θα ήθελα όπως και ο κύριος Ρικέ να πω πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση. Η ευρωπαϊκή κινητικότητα είναι ένα σημαντικό και επίκαιρο θέμα. Όλο και περισσότερο θα γίνεται επίκαιρο, διότι όλο και περισσότερες και πιο σημαντικές είναι οι προκλήσεις. Δεδομένου ότι όλοι οι πολίτες που ζουν σε ε, μεγάλες πόλεις έχουν προβλήματα κάθε μέρα περισσότερα. Παντού τα πάντα φρακάρουν. Όλοι έχουν πρόβλημα. Η Ευρώπη λοιπόν κάτι μπορεί να κάνει για να αμβλύνει αυτά τα προβλήματα. Και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξ της ομάδας μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν και να ασκήσουμε πιστεύω και περισσότερη πίεση στην Επιτροπή για να την υποχρεώσουμε να πάρει πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Δεν ξέρουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έκθεση της Επιτροπής. Ε, κάτι είχε λεχθεί για ένα δίκτυο βέλτιστων πρακτικών στις πόλεις. Πού βρίσκεται αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα λοιπόν, αν είναι παρόν κάποιος εκ μέρους της Επιτροπής, να μας ενημερώσει. Διότι ωραία είναι όλα αυτά τα οποία παριθμούνται εδώ ως ιδέες, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συνέση. Η κυρία Σάβισα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρόσπαχ για την εργασία που επιτέλεσε και όλα τα μέλη που κατέθεσαν τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας συμφωνεί με όλες τις τροπολογίες τις συμβιβαστικές στις οποίες και οι δικές μου ελήφθησαν υπόψη σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη κάποιες τροπολογίες που δεν έχουν κατά την άποψή μου θέση εδώ. Κατά την άποψή μας, κάποιες τις οποίες δεν υποστηρίζουμε είναι πολύ συγκεκριμένε ή πολύ λεπτομεριακές και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εδώ πρόκειται για μία γνωμοδότηση και για το μέλλον Ε, της ε, στα πλαίσια της πολιτικής συγγενής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Αστικό Περιβάλλον. Άρα δεν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ λεπτομεριακοί. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα πάντα. Βεβαίω πολλά προβλήματα απτώνται του αστικού Περιβάλλοντος. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και θέματα με τα οποία δεν συμφωνούμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μόνον ε, ε, αντίθετοι είμαστε με αυτές τις τροπολογίες που δεν υποστηρίζουμε, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να διηλύσουμε τον κόνοπα και να λύσουμε όλα τα προβλήματα των μεταφορών. Συμπερασματικά, πρέπει να πω ότι όπως και οι άλλες πολιτικές ομάδες και εμείς υποστηρίζουμε την έκθεση της κυρίας Ρόσπαχ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ για τους πράσινους. Ναι, πρόεδρε, να ευχαριστήσω την συγγετρία. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Οι συμβαστικέ προτάσεις που καταλήξαμε φυσικά θα τύχουν υποστήριξη από εμά. Ε, κάτι που είπε και η ίδια. για την ε, κατατμήματα ψηφοφορία να έχουμε 40% για τους ε, για τους σιδηροδρόμους, αλλά στο σημείο που έχουμε φτάσει νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε επιτύχει. Αλλά θέλω και μία διευκρίνηση για την τέταρτη, τον συμβαστικό, συμβαστική πρόταση D, για το mobility trains. Μήπως πρέπει να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, να πούμε ε, car sharing, car pooling, walking ε, κτλ. Δηλαδή όλα αυτά είναι μεταφορές, ένα είδος μεταφοράς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συμπληρώσουμε να στην συμβαστική πρόταση και αν μπορείτε θα θέλαμε την υποστήριξή σας εφόσον βεβαίως και η, η συγγήτρια το δέχεται αλλά και μετά όσα είπε ο κύριος Γκρός δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα αφού μας είπε ότι το 40% είναι εντάξει. Um, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Ρόσπαχ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έκανε. Και ενώ ο συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε βελτιώνει ορισμένες πιο ακραίες τροπολογίες τις οποίες είχαμε δει αρχικά, νομίζω ότι ο κ. Δίκα στα σχόλιά του υπογράμισε ε, το θέμα. Είπε ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά την κοινωτική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Περί αυτού πρόκειται. Πέραν από ε, την πολιτική, η πολιτική ε, σε αυτόν τον τομέα των μεταφορών, όπως είπαμε, είναι αρμοδιότητες των εθνικών κυβερνήσεων και πιο πολύ αρμοδιότητες των τοπικών αρχών. Και έτσι θα έπρεπε νομίζω να είναι. Δεν πρέπει στο δικό μας το επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο, να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε ε, στις προνομίες των ε, κρατών και των τοπικών αρχών που αναλαμβάνουν πολύ μεγάλη ευθύνη για τις τοπικές μεταφορές. Αυτό είναι το πρώτο. Η δεύτερη παρατήρηση που ελπίζω να είναι πιο θετική είναι ότι πράγματι θα ε, πιστεύω ότι ορισμένα μέλη τα οποία ορθά έθιξαν αυτό το θέμα, είναι ότι πρέπει να γίνει ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με αυτή την εκούσια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Μόνο θετική μπορεί να είναι. Αλλά θα ήθελα εδώ να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις που έγιναν και από άλλα μέλη. Ο κ. η υπενθύμησε ότι η Επιτροπή που να κάνει τούτο ή το άλλο. Δεν θέλουμε η Επιτροπή να κάνει οτιδήποτε, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι, όπως είπα, να αναλάβουν την ευθύνη οι αρμόδιοι υπεύθυνοι στα διοικητικά επίπεδα. Και ε, επίση τα σχόλια τα οποία έγιναν ε, είναι σωστά για ορισμένε τροπολογίε. Ελπίζω ο κ. Κράμερ θα με συγχωρήσει ε, ό,τι αφορά τη δική του τροπολογία και δεν νομίζω να μπορέσω να επηρεάσω αυτό το οποίο λέει. Αυτή είναι όμως η δική μου γνώμη. Καταλήγοντας, Πρόεδρε, τι λέτε, λέει ο ναι. Καταλήγοντας, Πρόεδρε, όπως είπα στην αρχή, οι συμβιβασμοί βελτιώνουν την έκθεση, πιστεύω, σε σχέση με τις αρχικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα αύριο. Ευχαριστώ. Mrs. Rosbach, do you Θέλετε να απαντήσετε, κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επί τη αρχή. έχω την ίδια άποψη με τον κύριο Μπράτμπορν και την κυρία Σάβησα. Έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Ε, Ω ε, δαν, μέλος από τη Δανία νομίζω ξέρω τι, είναι, μπορεί να πάει στραβά και τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ε, Γενικώ έχουμε πρόβλημα με την έκθεση. Χωρίς μικρόφωνο τα σχόλια του κύριου Κράμερ. Είναι δύσκολο όμως να μπούμε τόσο πολύ σε λεπτομέρειες και να προβλέψουμε τι γίνεται με τις μικρές πόλεις και τα λοιπά. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό για όλους μας να υπάρξει έτσι μια, ένας, μια κατανομή, ένας ε, διαμοιρασμός. Γιατί υπάρχουν πολλές καλές προτάσεις οι οποίες δεν είναι τόσο λεπτομερείς για το τι θα πρέπει να κάνουν ή μπορούν ή δικαιούνται να κάνουν οι περιφέρειες και οι πόλεις. Ε, Εντάξει, δεν θα... Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε τόσο πολλέ λεπτομέρειε. Νομίζω ότι ε, ξέρουμε όλοι που είναι το πρόβλημα. Και αυτή την ελευθερία θα πρέπει, αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το λύσουμε. Και οι ε, περιφέρειες και οι πόλεις ξέρουν ποια είναι τα προβλήματά τους. Να τους, το, να τους ρυθμίσουμε τώρα τις υποθέσεις τους τόσο λεπτομεριακά δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ίσως θα πρέπει να το αφήσουμε λίγο πιο ελεύθερο το σύστημα για να είναι και πιο πρακτικό. Ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή αύριο και η Επιτροπή Ρέτζιο θα ψηφίσει το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. TNT, διευρωπαϊκά δίκτυα, ανταλλαγή απόψε με την Κομισιόν. Θα πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Πάκε, ο οποίος δεν είναι εδώ. Οπότε, ας κάνουμε ένα δεκάλεπτο διαλυματάκι και θα ξανάρθουμε στις ε, παραπέντε για να ακούσουμε τον κύριο Δάκη. Okay, I'll restart the meeting. I'll... Να ξαναξεκινήσουμε. Θα έρθουν εκεί οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πακέ που θα μας παρουσιάσει. Νομίζω το σχέδιο απόφασης για την ε, ε, επιλογή των ε, διευρωπαϊκών δικτύων για το πολιετές πρόγραμμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω σήμερα τα αποτελέσματα της επιλογής των προγραμμάτων TNT, ε, των διευρωπαϊκών δικτύων για το 2010. Παρουσιάζουμε σήμερα λοιπόν ε, την επιλογή αυτή ε, στην Επιτροπή σας πριν από την παρουσίαση που θα γίνει για την ε, χρηματοπιστωτική ενίσχυση των προγραμμάτων TNT, όπου τα κράτη-μέλη θα ψηφίσουν για την επιλογή. Η συνάντηση αυτή θα γίνει αύριο και μετά ελπίζω ότι θα υπάρξει υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, οπότε να ξεκινήσει η συνήθις διαδικασία που θα είναι η γνωμοδότηση από το Κοινοβούλιο, αλλά ε, η Επιτροπή σας, ε, ως συνηθίζεται, είναι η πρώτη που θα λάβει γνώση των ε, αποτελεσμάτων της επιλογής. Έχουμε δύο προγράμματα εργασίας για το 2010 που εγκρίθηκαν από την Επιτροπολογία τον, την Άνοιξη. Ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Το ετήσιο έχει διάφορα στοιχεία τα οποία που, ε, θα αναφέρω παρόλο που δεν είναι το ουσιώδες της σημερινής ε, συνεδρίασης, είναι η, ε, τα 80 εκατομμύρια ευρώ που πάνε στο δίκτυο Μαργκερίτ, το οποίο ε, ιδρύθηκε το 2010. Μην με ρωτήσετε τίποτα για το Μαργκερίτ ακόμα, γιατί τώρα ξεκινά να δραστηριοποιείται αλλά και η, Επιτροπή, και η Τράπεζα συγγνώμη, Ευρωπαϊκών Επενδύσεων και το Μαργκερίτ θα κατασταλάξουν στο πώς ακριβώς θα γίνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο αυτό στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης, 50 ε, εκατομμύρια για, για το εργαλείο εγγύσεων δανειοδότησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Κομισιών για το LGTT η τράπεζα μας είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει επιπλέον 45 εκατομμύρια για το 2011. Οπότε όταν λάβαμε το αίτημα από την τράπεζα, λάβαμε και μια απόλυτα πλήρη το LGTT. Και βεβαίω, αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει, θα μπορούσαν οι συνάδελφοι από την τράπεζα να σας δώσουν μια παρουσίαση για το ποια είναι τα projects που διευκολύνονται και που χρηματοδοτούνται από το LGTT. Η βασική, το βασικό μας του προγράμματος εργασίας ήταν αυτό που συνήθως κάνουμε, το ετήσιο δηλαδή πρόγραμμα εργασίας για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών δικτύων. Έγιναν κάποιες ε, μελέτες και σε αυτό το ετήσιο πρόγραμμα, όπως το θυμάστε, προσθέσαμε δύο νέες προτεραιότητες. Μία να προετοιμάσουμε την, ε, τα προγράμματα TTT ε, και να διευκολύνουμε πιλωτικά προγράμματα με βάση και τις ε, ε, τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτέ ήταν οι δύο προτεραιότητε για το ε, πρόγραμμα εργασία μα το ετήσιο. Και θα σα πω και ποια προγράμματα προκύπτουν. Επίσης, μετά το, εκτός από το ετήσιο πρόγραμμα, είχαμε το πολιετέ για το 2011. Ε, για, το, για το 85 εκατομμύρια ευρώ για τους, ε, για, τις θαλάσσιες, στους διοδρόμους και το πολιετές πρόγραμμα για, τις, ε, για τους ποταμούς με 10 εκατομμύρια. Δεν θα σας κουράσω με τα συνήθη για το πώς γίνεται δηλαδή η Επιτροπή, πώς γίνεται η επιλογή. Η Επιτροπή σας το έχει ακούσει πολλές φορές. Βασιζόμαστε στην ποιότητα των προτάσεων που πρέπει να έχουν και την απαραίτητη τεκμηρίωση και μετά μπαίνουμε σε μια εις ανάλυση που μας, ε, για την οποία μας βοηθούν και εμπειρογνώμονες από, την, ε, από την φορέα για τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα προτινόμενα projects πάνε στην ε, Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αξιολογεί την προσθέμενη αξία τους. Η αξιολόγηση αυτή και η διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικές στις περισσότερες ε, τις περισσότερες φορές έχουμε πολύ περιγραφικές παρατηρήσεις. Έχουμε 3,5% περισσότερο, 3,5 φορές συγγνώμη, περισσότερες αιτήσει για ενίσχυση. Προσπαθούμε λοιπόν να επιλέξουμε τα προγράμματα που είναι τα πιο αποτελεσματικά, ειδικά σε ό,τι αφορά την καινοτομία και την ε, προσθέμενη αξία. Βέβαια αυτό είναι δύσκολο να γίνει γιατί σημαίνει ότι μπορούμε, μπορεί να απορρίψουμε ε, κάποια αρκετά καλά προγράμματα των οποίων όμως η προστιθέμενη αξία δεν είναι εξίσου υψηλή. Επίσης, Έχουμε δώσει μια μπροσούρα στην Επιτροπή σας ε, που έχει όλες τις ε, λεπτομέρειες για την υποβολή προτάσεων και την διαδικασία επιλογής και θα δείτε κάποια στατιστικά στοιχεία στην μπροσούρα αυτή για το ποια είναι τα προγράμματα που, που προτείνονται. Θα δείτε επίσης τον κατάλογο των projects που θα διατηρηθούν για την χρηματοδότηση και συμπεριλαμβάνουμε και έναν κατάλογο των ε, projects τα οποία δεν τα κατάφεραν. Θα έχετε λοιπόν και το αντίτυπο αυτό θα είναι και δημοσίως ε, διαθέσιμο βεβαίω, ώστε να έχετε μια γενική εικόνα πλήρη του καταλόγου που υπευλήθη κατά τη διάρκεια αυτή τη ε, υποβολή ενδιαφέροντος. Σύντομα, για, τους, ε, για τη θάλασσα και τους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους. Ο τρόπος αυτός ε, μεταφοράς ε, πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός. Μιλούμε επίσης για την εκνασιμότητα των αγαθών, γιατί το θέμα της διαχείρισης ε, είναι λιγότερο εδώ, για τις, για τις δηλαδή, σε σχέση με τις οδικές ή τις υδρονομικές μεταφορές. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Υπάρχουν πέντε προτάσεις και οι πέντε ήταν πολύ, καλές, ε, πολύ καλά προετοιμασμένες, με καλές συστάσεις ε, και επίσης ήταν λίγο κάτω από τον ε, προβλεπόμενο προπολογισμό. 7,1 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή θα δοθούν και 10 εκατομμύρια είχαμε διαθέσιμα. 2,9 λοιπόν δεν θα δοθούν. 2,9 εκατομμύρια. Θα υποστηριχτούν λοιπόν αυτά τα προγράμματα. Τώρα για τους ε, αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Θα θυμάστε ότι κάθε φορά ήταν δύσκολο να δώσουμε τα σωστά κονδύλια με βάση τις προτάσεις. Ήταν περιορισμένη η ποιότητά τους. Θα θυμάστε ότι λάβαμε υπόψη και την δυσκολία που έχουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα να υποστηρίξουν προγράμματα για τη θάλασσα και το πρόγραμμα εργασία για του αυτοκινητοδρόμου τη θάλασσα και αυτό που θέλαμε να επιτύχουμε ήταν ε, έτυχε αναθεώρηση. Έγιναν λοιπόν κάποιε αλλαγέ για να διευκολύνουν ε, την προετοιμασία των ε, projects και ειδικά των projects που αφορούν τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Υπάρχει ένας operator ε, στα πλαίσια του consortium που έχει αναλάβει την διαδικασία αυτή για την προετοιμασία των προγραμμάτων Επίσης διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή ώστε να επιτρέψουμε να γίνουν πιλωτικές μελέτες και με τις αλλαγές αυτές είχαμε μεγαλύτερη ε, επιτυχία, προτάθηκαν περισσότερα προγράμματα, 14 ε, επιλέξιμα εξετάστηκαν, 185 εκατομμύρια ευρώ ε, θα αποδοθούν και από αυτές τις 14 προτάσεις θα διατηρήσουμε τις 8, οι οποίες θα λάβουν 84,8 εκατομμυρία ευρώ. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον ενδεικτικό προπολογισμό που έχουμε για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. Και θα δείτε τα projects αυτά, τα οποία θα τύχουν χρηματοδότηση. Είναι στην σελίδα 14. Εκεί είναι ο κατάλογος των προγραμμάτων ε, για, τις για την πληροφόρηση και τις υπηρεσίες του... των ποταμών και στις... στη σελίδα 16 θα δείτε τα 8 προγράμματα που θα τύχουν ε, χρηματοδότησης για, τις... Ε, για τους αυτοκινηδρόμους της θάλασσας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι Νομίζουμε ότι είναι πιο χρήσιμο τώρα το σύστημα σε σχέση με παλαιότερα και για το βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το νότο. Στην προσούρα επίσης θα δείτε και ένα χάρτη, ο οποίος σας δίνει την γεωγραφική τοποθεσία αυτών των projects. Για το ετήσιο πρόγραμμα, Πρόεδρε, έχουμε τρία στοιχεία. Όλα αρκετά επιτυχή σε ό,τι αφορά τις προτάσεις. Πρώτη προτεραιότητά μας ήταν οι ε, απανθρακωμένες μεταφορές, δεύτερο ήταν η επιτάχυνση της εφαρμογής των TNT και τα τρίτο, το τρίτο ήταν οι εταιρικέ σχέσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είχαμε 3,4 φορές περισσότερες αιτήσει αυτή τη φορά, λάβαμε 58 προτάσεις, 34 προτάσεις μας, συνεστά μας, ε, μας έγιναν συστάσεις για να χρηματοδοτηθούν με 17,8 εκατομμύρια ευρώ, λίγο πάνω δηλαδή από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 77 ε, εκατομμύρια ευρώ, όχι 17, συγγνώμη, 77 ε, εκατομμύρια ήταν ο ενδεικτικό προπολογισμό, 77,8 ήταν η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν καλή η ε, καλό, καλή ισορροπία, 38% ε, από την χρηματοδότηση, 55% για τις μελέτες και ε, επικεντρωθήκαμε και σε, πολυ, και σε, πολλά, σε προτάσεις που περίχαν πολλά μοντέλα. Νομίζω λοιπόν ότι η γενική επιλογή των προγραμμάτων είναι αρκετά ευρεία. Βλέπετε στο, στην προσούρα ποια είναι τα προγράμματα που ξεκινούν από την ε, σελίδα 20 για την προτεραιότητα 1 και συνεχίζουν στην σελίδα 24 για την προτεραιότητα 2 μετά στη σελίδα 29 για την προτεραιότητα 3 για τα PPPs και υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος projects που ξεκινά στον, στην σελίδα 30. 3,4 λοιπόν παραπάνω η χρηματοδότηση χρειάστηκε, 3,4 φορές παραπάνω από τον διαθέσιμο προπολογισμό. Υπάρχει και μια εξήγηση για το τι καλύπτει το κάθε πρόγραμμα αυτά που έχουν διατηρηθεί για χρηματοδότηση και στα δεξιά ε, σημειώνουμε γιατί δεν έχουν ε, περάσει τα προγράμματα που δεν πέρασαν τελικά. Ε, ελπίζουμε να είναι χρήσιμη αυτή η μπροσούρα, ελπίζουμε να είναι, θέλαμε να είναι σύντομα τα κειμενάκια που περιλαμβάνονται, με πληροφορίες από την υπηρεσία, ώστε αν θέλετε, αν θέλετε βεβαίως λεπτομερέστερες ε, πληροφορίες, ευχαρίστως να σας τις δώσουμε είτε για τα προγράμματα που πέρασαν, τις εξετάσεις τους, είτε για αυτά που δεν πέρασαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Κάνσα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πακέ, για την ε, πρότασή σας και για τα έγγραφα τα οποία μας διανύματε. Κύριε Πρόεδρε, Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Διερωτώ πραγματικά πώς μπορούμε εμείς να εκφέρουμε άποψη για το έγγραφο αυτό το οποίο τώρα μόλις έφτασε στα χέρια μας. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο στη θέση μου για να μπορέσω να το μελετήσω. Είναι δύσκολα τα πράγματα λοιπόν. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μας έχουν αποστολή ε, νωρίτερα τα έγγραφα. Για του χρόνου ελπίζω ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας για να τα αναλύσουμε, να τα μελετήσουμε και να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το πολιετές. Αφενός έχουμε το ΡΙΣ και τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, για τις οποίες θα ήθελα να πω κάτι. Πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Ίσως κάνω λάθος, αλλά έχουμε διαθέσιμα 85 εκατομμύρια ευρώ και 14 ε, προγράμματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί έχουν εγκριθεί τα 8 από τα οποία 4 αφορούν τη Μεσόγειο με λίγα κονδύλια και τα υπόλοιπα την ε, περιοχή της Βαλτικής με πολύ περισσότερα κονδύλια. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της Μεσογείου. Διότι πρόκειται για μία θάλασσα την οποία πρέπει να ενισχύσουμε δεδομένου ότι εκεί έχουμε πλοία που φτάνουν από τις αναδυόμενες χώρες Και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα κριτήρια τα οποία έπρεπε να πληρεί κανείς για να υποβάλει αίτηση. Ποια είναι τα κριτήρια που υπερίσχυσαν για να εγκριθούν κάποια προγράμματα από κάποιες περιοχές. Εάν δεν συμμετάσχουν και οι χώρες της περιοχής ε, αν δεν συμμετάσχουν εκτός από τις ευρωπαϊκές ε, χώρες και οι χώρες της άλλης πλευράς ε, της ε, Μεσογείου και υπόλοιπες χώρες, τι κάνουμε. Στη Βαλτική βεβαίως έχουμε μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Η νότιος όμως Ευρώπη είναι διαφορετική υπάρχουν εμπορικές ε, συμφωνίες και σχέδια τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πολύ θελητική εξέλιξη για την ανάπτυξη της περιοχής, άρα και της Ευρώπης. Τον Οκτώβριο του 2009 στην Νάπολη είχαμε στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Δεν βλέπω όμως εδώ πέρα καμία αναφορά. Δεν βλέπω τίποτε. Επίσης, υπάρχει στο κεφάλαιο 9 ένα σχέδιο 2, 4 και 5 που αναφέρει ε, κάτι για την Αδριατική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία προοπτική ανάπτυξης για την περιοχή της Αδριατικής. Είναι λοιπόν σημαντικό να συμπεριληφθούν όλα τα σημαντικά σχέδια. Κάποια άλλη παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον, διότι μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρός. Ευχαριστώ κύριε Πακέ για την παρουσίασή σας. Βεβαίω, όπως είπε και ο συνάδελφος, τελευταία στιγμή πήραμε το έγγραφο, δεν μπορέσαμε να το διατρέξουμε, άρα δεν μπορώ να κάνω συγκεκριμένες παρατηρήσεις, αλλά θα πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, οι βουλευτές έχουν την δυνατότητα να δουν πιο εμπεριστατωμένες εκθέσεις ή κάποιες αξιολογήσεις που έκαναν οι εμπειρογνώμονες ή εάν υπάρξει ανάγκη τους ε, φακέλους κάποιον, κάποιον για να μπορέσουμε να ξέρουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Επίσης, αναφέρεστε στο ετήσιο πρόγραμμα του 2010 και αναρωτώ ποια είναι η σχέση μεταξύ του Μάρκο Πόλο και της πρώτης προτεραιότητας. Ποια είναι η σχέση ή υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Τελευταία ερώτηση εκ μέρους μου. Στον πρόλογο, στην εισαγωγή, αναφέρεται και άλλα κονδύλια. την Μαργκερίτ. Αλλά δεν βλέπουμε μετά να έχουν συμπεριληφθεί στο πακέτο. Άρα, πού θα πάνε όλες αυτές οι πιστώσεις. Θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας νέας έκθεσης. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες θα, πά, δοθούν σε άλλα σχέδια. Ευχαριστώ, κύριος Λοζιές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Λοιπόν, δεν θα κάνω άλλες μου παρατηρήσεις. Αλλά επιφυλασσόμεθα εκ μέρους της ομάδας για να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα μόνα που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι απογοητευτικό να βλέπουμε τι λέγεται για τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας. Επανειλημμένα είχαμε τονίσει ότι αυτό θα ελαφρύνει άλλους, άλλα μέσα μεταφορών, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψη επαρκώς οι παρατηρήσεις μας. Κρίμα. Μία άλλη ε, παρατήρηση. Ο κ. Σίμψον σίγουρα θα επανέλθει από αυτού. αναφέρουμε στον προγραμματισμό. Κύριο Σίμψον θα αναφερθεί ε, στη γνωμοδότηση με την Επιτροπή ΣΟΟ και θα μιλήσει για το χρονοδιάγραμμα των δημοσίων έργων και νομίζω ότι αυτό ανοίγει το δρόμο για ένα προγραμματισμό που συζητείται τώρα στην Επιτροπή, δηλαδή ότι πρέπει να προβλέπετε περισσότερος χρόνος από ό,τι έχουμε σήμερα, διότι είναι πέντε χρόνια συν πέντε αυτή τη στιγμή. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν δέκα χρόνια κάτι το οποίο επιθυμούμε. Καλό θα ήταν τα έγγραφα να φάνουν έγκαιρα. Ευχαριστώ. Ähm, Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Εάν λάβουμε τόσο σύντομα ένα, πρόβλημα, ένα πρόγραμμα, δεν γίνεται να αξιολογήσουμε την, την ποιότητά του. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με βάση δηλαδή και επιστημονικές μελέτες που θα θέλαμε, γιατί ούτως ή άλλως κάποια προγράμματα είναι καλύτερα. Οπότε καλό θα ήταν ε, να τα λαμβάνουμε λίγο πιο έγκαιρα, για να μπορούμε και εμείς εδώ να κάνουμε μια καλή συζήτηση, να θέτουμε τα ερωτήματά μας, να παίρνουμε τις απαντήσεις μας, για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Γιατί αλλιώς ε, θα είναι σαν να συμμετέχουμε ιονοί και δεν νομίζω ότι αυτό το θέλουμε και λόγω των, της σημασίας που έχουν τα δίκτυα αυτά και λόγω των ποσών για τα οποία μιλούμε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Σε αυτές τις συζητήσεις θέλουμε να λαμβάνουμε έγκαιρα τα έγγραφα. Ε, είναι ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει. Μόνο έτσι ακροθυγός μπορώ να θέξω κάποια πράγματα. Γιατί δεν είχα και το χρόνο να τα μελετήσω. Ε, μιλήσατε για την προετοιμασία των ε, συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Τι ακριβώς σημαίνει όμως αυτό γιατί είναι σημαντικό σημείο. Δεύτερον, η ιστορία αυτή με τα, τα προγράμματα πληροφόρησης για τους ποταμούς και τα σχετικά συστήματα. Εδώ οι παρατηρήσεις μου όταν το αποφασίσαμε το πρόγραμμα αυτό ε, ήταν, είχε να κάνει με την διαλειτουργικότητα. Το ξαναθέτω. Αυτά τα συστήματα που, για τα οποία μιλούμε εδώ είναι διαλειτουργικά ή είναι μονοπωλιακά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουμε όσοι ε, κυκλοφορούν σε ποταμούς ε, να μην αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ένα, το ένα ή το άλλο σύστημα, να μπορούν τα συστήματα αυτά να είναι ευέλικτα και διαλειτουργικά. Τρίτο σημείο. Είπατε, αυτοί που είναι, αυτά που είναι αρκετά καλά. Τι θα πει αρκετά καλά. Ε, μου χτύπησε λίγο περίεργα στα αυτιά η λέξη αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς είναι το quite okay που είπατε, το αρκετό καλό. Δηλαδή με βάση τα κριτήρια τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα ήθελα να μου πείτε. Με ενδιαφέρει. Και επίσης με εξέπληξε λίγο. Γιατί το Malpensa είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόγραμμα. δεν συνδέονται τα δύο ε, τέρμιναλ, οι δύο αεροσταθμοί του αεροδρομίου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα λαθασμένου σχεδιασμού. Και θα ήθελα και μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Δηλαδή, να μας δώσει μια ημερομηνία, να μελετήσουμε το έγγραφο λεπτομερώς και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και λεπτομερώς. Είδα πια τις απορρίψεις που έχετε κάνει αλλά θα ήθελα κάποιες ακόμη πληροφορίες. Γιατί κάποια <coughs> έτυχαν εξέταση από εξωτερικούς ε, ελεγκτές και κάποια όχι. Παρακαλώ να μην ε, παίρνετε περισσότερο χρόνο, ώστε και η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να απαντήσει. Ο κ. Δικέ. Πρόεδρε, πρώτη παρατήρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πακέ για την παρουσίασή του. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, δεν έχουμε αρκετό χρόνο, Λαμβάνοντα υπόψη την πολυπλοκότητα αυτού του θέματος. Αλλά θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, και ελπίζω ο κύριος Πακέ θα μου το επιτρέψει, να θέσω ένα ερώτημα. Κάτι το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Πριν από αυτά τα προγράμματα, η Επιτροπή αναθεώρησε όλα τα στοιχεία του προπολογισμού για τον ε, προπολογισμό του, του RTOT και εδώ ένα θέμα ε, είναι σημαντικό για μένα, είναι το μόνο ε, ποτάμιο πρόγραμμα, ένα δύσκολο πρόγραμμα για να στηθεί, διότι γίνεται η χρηματοδότηση από πολλούς και τέσσερις χώρες συγκεκριμένα ευρωπαϊκές παρά την κρίση και βλέπω τη στιγμή που έχει εγκριθεί ο προπολογισμό, η Ευρώπη, η Επιτροπή αποφασίζουν να διαγράψουν 40 εκατομμύρια στη χρηματοδότηση. Υπήρχε ένα έλλειμμα 60 εκατομμυρίων στη χρηματοδότηση που μόλι είχε καλυφθεί και τώρα βγάζουμε 40 δισεκατομμύρια. Μου πενθυμίζει ότι όταν δίνω ένα λουκάνικο, ένα ε, σαλάμι στον ε, σκύλο μου και ε, πηδάει για να το πιάσει και το του τραβάω. Το ίδιο συμβαίνει εδώ. Δεν μπορεί λοιπόν να το σκεφτεί αυτό η Επιτροπή. Είναι λογικό σε αυτό το θέμα ε, να γίνεται αναθεώρηση δημοσιονομική και να υπάρξει τέτοια περικοπή ε, του κονδυλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα πάλι. Λυπούμε που Πρέπει έτσι τρέχοντας να το δούμε αυτό το κείμενο. Θα πω απλώς ότι πολλά μικρά προγράμματα μπορούν να κάνουν ένα μεγάλο. Και υπάρχουν τέτοια προγράμματα στην, στην ε, μπροσούρα σας. και δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς τα έχετε, ε, τα έχετε ακριβώς συνδυάσει. Ας πούμε τα, τα προγράμματα μεταφοράς από δικές σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες μεταφορές. Είναι αξιόλογα προγράμματα, τα οποία όμως δεν τα βλέπω εδώ να έχουν τεθεί ως προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι συμβαίνει με τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας. Ήδη είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα για τη Μαύρη Θάλασσα και για τη Μεσόγειο αλλά δεν τα βλέπω εδώ. Για ποιο λόγο. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ληφθεί υπόψη δεόντως αυτό το πρόβλημα. Αναφορικά με το πρόγραμμα 2010 έχω ένα ερώτημα. Κανένα ρουμανικό πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί ούτε απορριφθεί. Γενικά δεν υπάρχουν αιτήσει από τις νέες χώρες. Τι πρέπει να γίνει για να απαντήσουμε σε αυτά τα θέματα. Ε, είμαι σίγουρος αν ε, ε, ήταν δικό σας θέμα και δεν υπήρχε πρόβλημα χρημάτων, θα λέγατε ναι σε όλα τα προγράμματα. Ο πραγματικός κόσμος είναι διαφορετικός όμως. Το λόγο έχετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία σας δώσαμε τα έγγραφα τα τα λάβατε μαζί με τα κράτη-μέλη, συνεπώς ε, θα έχουμε αντίδραση φαντάζομαι αύριο από τους συναδέλφους και τις εθνικές διοικήσεις. Ε, ε, θα φροντίσουμε την επόμενη φορά να λάβετε τα έγγραφα έγκαιρα. Πάλι όμως, αν θέλετε επιπλέον πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας. Μπορούμε να σας πούμε ποια προγράμματα έχουν γίνει δεκτά ή όχι. Η εξωτερική εξολόγηση αναφέρεται για τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί. Για όλα εκείνα τα οποία έχουν εγκριθεί, η εξωτερική αξιολόγηση υπήρξε θετική, γι' αυτό και δεν το αναφέρεται. Στι περιπτώσει όμω των προγραμμάτων που απορρίπτονται, υπάρχουν ορισμένε περιπτώσει όπου η εξωτερική εξολόγηση είπε ναι, μεν, αλλά η Επιτροπή τελικά ε, επειδή έπρεπε να κάνει επιλογές, ε, απέριψε ορισμένα. Και σε ορισμένε περιπτώσει, ε, όταν οι εξολογητές μας είπαν να μην προχωρήσουμε, δεν προχωρήσαμε, αλλά τα εξηγούμε. Μπορούμε, αν θέλετε, να σα δώσουμε περισσότερε πληροφορίε, όπω σα είπα, αν το ζητήσετε. Τώρα, σχετικά με του αυτοκινητόδρομο τη θάλασσα. Ναι, δεν ζητήθηκε τίποτα από τη Ρουμανία και γενικά λίγα προγράμματα ε, ζητήσαν για τις, ε, αυτοκινητόδρομους της θάλασσας και λίγα από τα νέα κράτη. Αυτό είναι απογοητευτικό επειδή το ετήσιμο πρόγραμμα ε, σε μεγάλο βαθμό είχε αντικείμενο να ετοιμάσει ε, το πρόγραμμα κατόπιν ετήσεω των χωρών. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε με τι διοικήσει αύριο για να δούμε για ποιο λόγο αυτό συνέβη. Επίση, μα ανησυχεί το γεγονό ότι μία από τι προθέσει ότι μία από τι προθεσει όσον αφορά το μελλοντικό πλαίσιο χρηματοδοτηση είναι καλύτερη διάρθρωση μεταξύ ε, των ταμείων χρηματοδότησης και ελπίζουμε ότι το 2011 και 2012 θα δημιουργήσουμε το project pipeline για το μελλοντικό πλαίσιο συνοχής. Πράγματι πρέπει να φροντίσουμε ότι υπάρχουν τα προγράμματα και το 2010 δεν είχαμε σχεδόν κανένα. Ε, αυτό απασχολεί και εμάς. Τώρα, όσον αφορά την ε, ε, Μεσόγειο ε, και τα, τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, έχουμε τέσσερα προγράμματα, τα καλύτερα που είχαμε. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος, θα έλεγα. Επίσης, στο ετήσιο πρόγραμμα έχουμε ένα project που ονομάζεται Adriatic Gateway, που συνδέει το, τη Βόρεια Μεσόγειο με το σύστημα χερσαίων μεταφορών, ώστε να υπάρχει σύνδεση ε, με, ε, μεταξύ των μεταφορικών μέσων. Τώρα, όσον αφορά ορισμένες χώρες, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε projects ε, που πηγαίνουν στην Αφρική ή στην Τουρκία, για παράδειγμα, σε περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό δεν προβλέπεται. Αλλά στα πλαίσια του, της περιφερειακής μας συνεργασίας υποστηρίζουμε περίπου έξι επιπλέον projects για του αυτοκινητόδρομου τη θάλασσα Υπήρχαν λιγότερα χρήματα, αλλά υπάρχουν ορισμένα project για τις εξωτερικές, ε, για το, στα πλαίσια του προγράμματο των εξωτερικών σχέσεων μεταξύ Μεσογείου και Αφρική. Η σχέση μεταξύ προτεραιότητα 1 και Μάρκο Πόλε με δύο λόγια είναι υπηρεσίε αφενό και υποδομέ αφετέρου αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά αν θέλετε και ε, το θέμα του, της καλύτερης ενσωμάτησης μεταξύ Μαρκοπόλο και ΤΕΝΤΗ ε, των διευρωπαϊκών δικτύων πέραν των αυτοκινητοδρόμων της θαλάσσης. Εδώ συζητούμε στην Επιτροπή για ένα ενοποιημένο πλαίσιο χρηματοδότησης για τις ε, μεταφορές και το 2011 και 2012 θα προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ Μαρκοπόλο και ΤΕΝΤΗ και στο προγραμματισμό για να υπάρξει η μέγιστη συνέργεια και να μην υπάρξουν προβλήματα ε, όπως εκείνα τα οποία θίξατε. Για τη Μαργκορίτ και την NGTT, η Μαργκορίτ είχαμε 80 εκατομμύρια για το Equity Fund. Μόλις ξεκίνησε τώρα και προτείνω το 2011 με τη διαχείριση του Μαργκορίτ και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δούμε, να κάνουν απολογισμό ε, για το τι έκαναν μέχρι εκείνη την εποχή. Ακόμα δεν υπάρχουν προτάσεις χρηματοδότησης. Νομίζω ότι θα προκύψουν το 2011. Φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν και projects στο TEN-T για να δικαιολογηθεί η χρηματοδότησή του. Για το NGTT Εκεί υπάρχει ένα project καθοδόν, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά όπως σας είπα, η τράπεζα είναι θετική όσον αφορά το LGTT και θα ζητήσουμε 45 εκατομμύρια επιπλέον για το LGTT και αυτό θα είναι στο ετήσιο πρόγραμμα του χρόνου και το ετήσιο πρόγραμμα φυσικά υπόκειται στην επιτροπολογία θα σας ενημερώσουμε σχετικά και τότε προτείνω να γίνει μια παρουσίαση ε, για το project του NTCC και μια γενική συζήτηση ε, που θα περιλαμβάνει και τη Μαργκορίτη. Η Μαργκορίτη είναι με διαφορετική περίπτωση γιατί είναι ένα private equity fund που έχει διαφορετική δομή ε, δίκησης. Τώρα, οι συνδυασμένες μεταφορές δεν είναι επικεφαλή στη λίστα των προτεραιοτήτων. Στο ετήσιο πρόγραμμα δώσαμε μεγάλη σημασία στους σιδηροδρόμους και στις πλωτές οδούς και στους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας. Ειλικρινά δεν υπάρχουν άλλα projects, άλλες μορφές project. Αυτή είναι μια πολιτική προτεραιότητα την οποία βλέπουμε και στα projects τα οποία παρουσιάστηκαν για ε, τις ΔΙΤ τώρα ε, στηρίζουμε τρεις μελέτες. Η, ιδέα στο πρόγραμμα εργασίας ήταν η εξής. Αυτές οι τρεις μελέτες θα αποτελέσουν τη βάση ειδικά project. Το ένα στην Ολλανδία, το λιμάνι του Άμστερνταμ, ένα project σιδηροδρομικό στη Φινλανδία και κατόπιν υπάρχει ένα project πάλι συνδρομικό στην Πορτογαλία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια των ΣΔΙΤ είναι να υποστηρίζουμε τα project τα οποία είναι καινοτόμα. Όχι χαρακτηριστικές οδικές ε, πρωτοβουλίες που έχουν συνηθίσει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Πήραμε τρία μάλλον δύσκολα project που θα είναι καλής ποιότητας και ελπίζουμε να βοηθήσουμε ε, καινοτόμα προγράμματα ΣΔΙΤ ε, στον τομέα των σιδηροδρομικών και θαλασσίων ε, μεταφορών. Μαλπένσα τώρα. Έχει σχέση με το σιδηροδρομικό σύστημα εδώ. Μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής TNT σήμερα και μελλοντικά είναι να συνδέσει τα αεροδρόμια με ε, σειρμούς μεγάλης ταχύτητος και το αντικείμενό μας είναι να επιτρέψουμε και να ετοιμάσουμε την σύνδεση του αεροδρομίου με ταχείες. Ε, ε, δεν ε, τώρα, όσον αφορά τους κινδύνους των μονοπωλίων και την διαπιχειρησιακότητα, διαλειτουργικότητα, υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των projects, αλλά με τα χαράς να το συζητήσω μαζί σας, διότι δεν το είχα απόψη μου. Ο κύριος Ρικέ, θα σας απαντήσω και εσάς το ερώτημά σας αφορούσε περισσότερο την ενδιάμεση αναθεώρηση που παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στην Επιτροπή σας. Θα θυμάστε ότι η ισορροπία που είχε βρεθεί από την Επιτροπή ήταν να εξασφαλίσει πράγματι μια επέκταση δύο ετών στο project, το οποίο είχε καθυστερήσει στην υλοποίησή του, μεταξύ των οποίων και το ΣΕΝΕΣΚΟ, αλλά πέρα από το 2015 οι δραστηριότητες δεν θα υποστηρίζονταν πλέον επειδή από το 2013-2014 θα υπάρξουν άλλε χρηματοδοτήσεις και πρέπει να βρούμε την καλή ισορροπία μεταξύ των projects και της χρήση των περιορισμένων κονδυλίων στα πρόγραμματα Dante. Επίσης, ήταν σημαντικό για μα να εξασφαλίσουμε στα πλαίσια της ΕΝΕΣΚΟ ή άλλου project, της Fem Health που ξεπερνούσε το έτος 2015, ότι αυτές οι περικοπές δεν θα έθεταν σε κίνδυνο το project και τώρα συζητούμε με τις ε, αρμόδιες αρχές της Δανίας και της Γαλλίας ώστε να μην υπάρξουν αυτές οι περικοπές. Και τώρα από πλευρά ΕΝΕΣΚΟ η διοίκηση των πλωτών οδών της Γαλλίας προσπαθεί να μας καταδείξει ότι ίσως ίσως βιαστήκαμε εφόσον αυτές οι, προτεραιότητες, οι ξεπερνούσαν το 2015 Εάν ε, περιορίζονταν το 2013-2014, η περικοπή θα έπρεπε να επανεξεταστεί υπό το φως των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει. Ευχαριστώ. Καλό να σχολιάσετε σε συντομία γιατί βλέπω ότι ε, και άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Να είσαστε πολύ σύντομος παρακαλώ. Δεν θέλω να σχολιάσω, όχι, απλά και μόνον ήθελα να διορθώσω κάτι το οποίο είπα πρωτήτερα, διότι δεν, το δεν ερμηνεύτηκε σωστά. Δεν σας είχα πει ότι θα έπρεπε οι, τα λιμάνια της Αφρικής ή της Ασίας να εμπλακούν, αλλά έλεγα ότι η μέθοδος αξιολόγησης ε, σε σχέση με τη Βαλτική που περιβάλλεται από ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή υπάρχουν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες γύρω από τη Βαλτική και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ε, που θίγονται. Ίσως λοιπόν η μέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να επανεξεταστεί. Τώρα για το project Marguerite που αρχίσαμε να χρηματοδοτούμε, καλό θα ήταν να έχουμε ορισμένα στοιχεία, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Πακέ ή όχι. Δεν, νομίζω δεν κατάλαβα την τελευταία ερώτηση. Για το Marguerite ήταν τελικά. Για τη Marguerite, σε τι αναφερθήκατε. Για το Marguerite, σας κατάλαβα ή όχι, δεν ξέρω. Αναφερόσασταν στο Μαργκορίτ ή όχι. Μαργκορίτ, think. Ναι, για το Μαργκορίτ ήταν. Για το Μαργκορίτ. Λοιπόν, είπα η Μαργκορίτ είναι ένα private equity fund που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους χρηματοπιστωτικούς ε, οργανισμούς και προτείνω να ζητήσουμε στη διοίκηση της Μαργκορίτ αν θέλει να έρθει σε αυτή την Επιτροπή και να κάνει μια παρουσίαση για τη λειτουργία της. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό και για σας αλλά και για τη Μαργκορίτ πιστεύω. Αυτό με διευκολύνει στο πρόγραμμά μου, το χρονοδιάγραμμά μου των επομένων 12 μηνών. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ας έλθουμε ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών. Λύεται η συνεδρίαση και τώρα θα έχουμε τους συντονιστές.